liebe Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Τουλάχιστον αυτοί που είναι εδώ παρόντες. Ερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε κάποιες τροποποιήσεις για την ημερήσια διάταξη. Εδώ βλέπω να υπάρχουν όμως κάποιες αλλαγές, κάποιες αιτήσει αλλαγών γιατί είναι άλλοι συνάδελφοι που έχουν άλλες συνεδριάσεις ή άλλα κολλήματα παράλληλα. Θα προσπαθήσω στο μέλλον να περιορίσω αυτές τις αλλαγές στο ελάχιστο, γιατί είχαμε ήδη μεγάλες δυσκολίες να αλλάξουμε την αλληλουχία των σημείων. Αν συμφωνείτε λοιπόν το σημείο 15 μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μετά το σημείο 7 σήμερα το πρωί, το δε σημείο 8, στις 4 η ώρα να το αναβάλουμε το απόγευμα θα ξεκινήσουμε με τα σημεία 9 και 10 και το σημείο 17 θα το εξετάσουμε μετά από το σημείο 11 σήμερα το απόγευμα. Έχετε αντιρρήσεις για αυτή τη διαδικασία. Είσαστε όλοι ενθουσιασμένοι. Θαυμάσαι. Πώς. Όλοι συμφωνούν. Εντάξει. Φαντάζομαι ότι οι εμπλεκόμενοι με αυτές τις αλλαγές έχουν πληροφορηθεί και θα είναι εδώ και η μόνη μου παρατήρηση για το σημείο 2 είναι ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα, στην διαχείριση του χρόνου για να προλάβουμε όλα αυτά τα θέματα. Αύριο το απόγευμα δεν θα έχουμε συνεδρίαση, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα δράσουμε με αυτοπιθαρχία για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε τον απαραίτητο χρόνο. Δεν έχω λοιπόν τίποτα να σας ανακοινώσω. Πάμε στο σημείο 3 λοιπόν. Χαιρετίζω τον καθηγητή κύριο Ρίτσελ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την αξιολόγηση του έκτου προγράμματος πλαισίου. Φυσικά έχει φέρει και μια παρουσίαση την οποία θα μας κάνει. Η έκθεσή του έχει συμπληρωθεί τον ε, Φεβρουάριο του 2009 και είναι επικεφαλής της ομάδας εμπειρογνωμόνων και Πιστεύω ότι μετά από την παρουσίασή του θα έχουμε καιρό για να, για να ανταλλάξουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Κύριε θα σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρόιλ. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω το αποτέλεσμα των εργασιών μας για μια αξιολόγηση του έκτου προγράμματος πλαισίου. Φυσικά έχει ε, εκπνεύσει το, έχετε περατωθεί το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ποια είναι τα προϊόντα αυτού του έκτου προγράμματος πλαισίου και να αντλήσουμε συμπεράσματα εν ώψη του όκτου προγράμματος πλαισίου. Είχε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτή η αξιολόγηση γιατί για πρώτη φορά προβήκαμε σε μια συνολική αξιολόγηση ενός προγράμματος πλαισίου. Στο παρελθόν είχαμε μονάχα αποσπασματικές αξιολογήσεις σε διαφορετικές ε, χρονικές στιγμές. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Δεύτερον, είναι η πρώτη φορά που ένα πρόγραμμα πλαίσιο έχει σχεδιαστεί για να επιτύχει μια σειρά πολιτικών στόχων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των στόχων της Λισαβόνας, της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. Αυτή ήταν η στόχη του έκτου προγράμματος πλαισίου και αυτό ήταν κάτι το καινοτόμο. Επομένως, η ομάδα αξιολόγησης ήταν πολύ μορφή και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον και θετικό ότι είχαμε εμπειρογνώμονες από διάφορες προελεύσεις οι οποίοι αντιμετώπισαν την αξιολόγηση αυτού του εγώ θα σταθώ τώρα σε δύο μονάχα προβλήματα, τα οποία εμένα μου φάνηκα ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικά σε ό,τι αφορά την διεξαγωγή του προγράμματος αυτού, πλαισίου και έχουν να μας δώσουν διδάγματα για την οργάνωση ενός προγράμματος πλαισίου στο μέλλον. Ένα από τα προβλήματα ήταν τα διοικητικά προβλήματα και ένα άλλο πρόβλημα ε, άλλα προβλήματα επιμέρους θα αναφέρω στην έκθεση. Το πιο σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαμε ήταν ότι καταρχήν θα έπρεπε να δούμε στην αξιολόγησή μας την πτυχή της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής Λισαβόνας. Ο στόχος, όπως αναφερόταν, ήταν να ενισχύσει την ε, επιστημονική βάση της βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενθαρρύνει τη βιομηχανία να είναι πιο ανταγωνιστική με το να παροτρύνει και άλλες ερευνητικέ προσπάθειες που είναι απαραίτητες από άλλα ε, κεφάλαια της συνθήκης, συγκεκριμένα το άρθρο 163. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο λοιπόν. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε επομένω ότι η γενική, η γενική λογική του προγράμματος πλαισίου να περιλαμβάνει υποστόχους και υπο που να μπορούμε να τους αξιολογήσουμε. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Εμείς είδαμε ότι από τον κύριο στόχο περάσαμε σε υπο, επιμέρους στόχους και εκεί υπήρξε ένα άλμα ή ένα χάσμα γιατί αυτοί οι επιμέρους στόχοι δεν ήταν αμέσα συνδεδεμένοι με τον ε, γενικό στόχο. Επομένω, μα ενδιαφέρει να ξέρουμε κατά πόσο αυτή η επιμέρου στόχη ήταν λογική, ήταν επιτεύξιμη και ήταν χρονικά καθορισμένη με σωστό, με σωστό τρόπο. Υπήρχαν τώρα υποστόχοι, όπως παραδείγματος χάρη, η πρόθεση της κινητικότητας των ε, ερευνητών. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ποσοτικοποιήσιμο και μπορεί κανείς να το μετρήσει. Ή επίσης η επιση η κοινών υποδομών. Προφανώς μπορούμε να δούμε ποιες υποδομές δημιουργήθηκαν, πόσες και ποιες και επίσης το να υπάρχουν κοινά πρότυπα για την ευρύτερη ασφαλή χρήση ραδιενεργών υλικών. Η Κομισιόν όμως θα πρέπει να σκεφτεί καλύτερα στο πλαίσια του όκτου ε, προγράμματος πλαισίου για υποστόχους όπως το να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας είναι δύσκολο να πει κανεί τι προωθεί και τι δεν προωθεί αυτή την ανάπτυξη, πώς θα αντιμετωπίσουμε την, τα δύναμα σημεία τη ευρωπαϊκή έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία. Είναι απαραίτητο λοιπόν οι επιμέρου στόχοι να έχουν διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν πράγματι να καταμετρηθούν και να αξιολογηθούν. Ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, και αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα γενικά μέσα στην συστηματική των ε, προγραμμάτων πλαισίου, είναι το θέμα της διοίκησης και της διαχείρισης αυτών των προγραμμάτων. Έχει αναφερθεί πολλές φορές το θέμα της ε, απλοποίησης και εμείς θεωρήσαμε καταρχήν ότι για τα θέματα διοίκησης και διαχείρισης δεν μπορούν τα πράγματα να προχωρήσουν. Χρειάζεται να υπάρξει μια συστηματική αλλαγή σε σχέση με τα διοικητικά θέματα. Εμείς βλέπουμε ότι η διοικητική αυτή, το διοικητικό άχθος το οποίο συνοδεύει αυτά τα προγράμματα ουσιαστικά στρέφεται κατά των Βρυξελών, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει ότι θα απλοποιηθεί το σύστημα αυτό, ώστε και οι ίδιοι οι βιομηχανικοί κύκλοι να θεωρήσουν ελκυστικά αυτά τα προγράμματα που περιέχονται στο πρόγραμμα πλαίσιο, αλλιώς θα έχουμε προβλήματα και αλλιώς δεν θα υπάρξει εκμετάλλευση αυτών των ευκαιριών από τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό θέλω να τονίσω την ανάγκη μιας σημαντικής απλοποίησης. Ένα άλλο πρόβλημα, όχι γενικό αλλά σε ορισμένα κράτη-μέλη, υπήρχαν πολλά κράτη τα οποία χρειάστηκαν αρκετό χρόνο για να καταλάβουν πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Κάτι όμως το οποίο δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι ότι τα προγράμματα πλαισίου πλαίσιο δεν δημιουργούνται μονάχα προ όφελο των επιστημόνων και των ερευνητών, αλλά και για τη βιομηχανία. Γιατί είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε συμμετοχή της ε, βιομηχανίας. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχει επαρκή συμμετοχή, μάλλον μειώνει τη συμμετοχή της βιομηχανίας και ένας από τους λόγους είναι ακριβώς το διοικητικό άχθος. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Για να συναυθεί μία σύμβαση χρειάζονται σε 75% των περιπτώσεων 450 ε, μέρες, δηλαδή σχεδόν 1,5 χρόνος. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο για τις περισσότερες βιομηχανίες. Δεν μπορεί κανείς να περιμένει 1,5 χρόνο για να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού και να έχουμε εδώ μια αποφασιστική αλλαγή. Βλέπετε επίσης ορισμένες προτάσεις οποίες έχουμε διατυπώσει. Καταρχήν μια εκβάθρον αναθεώρηση σε σχέση με την οτροπία που διέπει το σύστημα, η οποία πρέπει να ξεκινήσει τώρα ήδη η Κομισιόν μόνη της δεν μπορεί να το αποφασίσει. Πρέπει να υπάρξει και υποστήριξη από τα κράτη-μέλη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να φύγουμε από ένα σύστημα που περιέχει υπερβολικούς ελέγχους. <clears throat> Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη τα οποία έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά την διαχείριση των προγραμμάτων αυτού του είδους και έχουν απλοποιήσει πολύ τις διαδικασίες τους. Θα πρέπει οι Βρυξέλλες να ακολουθούν μια διαδικασία η οποία να είναι πραγματικά απλή, τόσο απλή όσο η απλούστερη διαδικασία που ισχύει στα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αυτονομία και ευκαμψία για τα κονσόρσια τα οποία συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, να υπάρξει μείωση του χρόνου μέχρι την ε, υπογραφή ενός μιας σύμβασης, 200 μέρες το πολύ, <clears throat> για να, για να τελειώσει αυτή η διαδικασία και επίσης να υπάρξει κάποια ενοποίηση μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του προγράμματος πλαίσιο και επίσης οι εκτελεστικοί φορείς μπορούν να έχουν μια θετική εξέλιξη αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε οι εκτελεστικοί αυτοί φορείς να μην κινούνται ανεξάρτητα από τις γενικές διευθύνσεις της Κομισιόν σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα, αλλά αντίθετα να συνεργάζονται. Αυτά είναι τα βασικά σημεία κριτικής που θέλουμε να διατυπώσουμε σε σχέση με το πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά από την άλλη μεριά είδαμε ότι υπήρχαν και πολλές θετικές πτυχές στο πρόγραμμα πλαίσιο. Διαπιστώσαμε, αντίθετα από την άποψη που έχουν ορισμένοι, ότι οι άριστοι ερευνητές και τα άριστα σχέδια έχουν περιληφθεί στο πρόγραμμα αυτό, είχαν περιληφθεί στο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν είναι ελκυστικά αυτά τα προγράμματα και συμμετέχουν μονάχα δευτεροκλασάτη επιστήμονες. Είχαμε βραβεία Νόμπελ τα οποία συμμετέσχαν. Δεύτερον, το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο έπαιξε ένα καταλητικό ρόλο στο να υπάρξει καλύτερη διαδικτύωση των ερευνητικών ιδρυμάτων, να αυξηθεί επίσης η, η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η, μέσω του προγραμμάτος πλαισίου υπήρξε μια τεράστια επιτυχία. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό μήνυμα το οποίο μπορώ να σας δώσω και συζητήσαμε πάρα πολύ για το αν υπάρχει κάποια αναλλακτική επιλογή εναντί του προγράμματος πλαισίου, καταλήξαμε η Επιτροπή Αξιολόγηση ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική ε, επιλογή η οποία θα μπορούν να είναι τόσο επιτυχής όσο το πρόγραμμα πλαίσιο. Είναι σαφές λοιπόν ότι είναι απαραίτητο ένα τέτοιο πρόγραμμα πλαίσιο, βέβαια με διαφορετική διάρθρωση, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό εργαλείο που θα προωθήσει την έρευνα και τη βιομηχανία. Συστάσεις. Κοιτάμε λιγάκι τώρα προς το μέλλον, το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο και τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να τονίσουμε ότι το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να εστιάζεται περισσότερο στη συνεργασία της βιομηχανίας με την έρευνα και την επιστήμη. Πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό και οι επιστήμονες τείνουν να βλέπουν το πρόγραμμα πλαίσιο σαν κάτι το οποίο θα τους δώσει χρήματα απλώς. Αλλά αν δεν υπάρχει σύνδεση με την βιομηχανία δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ε, το, νόημα λοιπόν του προγράμματος πλαίσιο είναι να ενισχύσει τους δεσμούς της ε, επιστήμης και της έρευνας με τη βιομηχανία. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε τη συμμετοχή της βιομηχανίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεύτερον, το σχήμα NEST. Θέλουμε να έχουμε προγράμματα τα οποία είναι διαδικτυωμένα μεταξύ τους θα ήταν λάθος να έχουμε μονάχα μεμονωμένα προγράμματα. Πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία στο 8ο πλαίσιο πρόγραμμα πλαίσιο και να θέσουμε σαν πρώτη προτεραιότητα τη συνεργασία και όχι μοναχά να προωθούμε μεμονωμένα προγράμματα. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις υποδομές δεν είναι απαραίτητο μονάχα να δημιουργήσουμε νέε υποδομέ, αλλά και να τι διατηρήσουμε, να τι συντηρήσουμε επίση. Και εδώ χρειάζεται μια κλίση προ την Κομισιόν για περαιτέρω χρηματοδότηση. Επίση, η εξασφάλιση ισότητα των φύλων, και αυτό ήταν κάτι το οποίο το αντιμετωπίσαμε. Υπάρχουν και θετικά και αρνητικά σημεία. Η Κομισιόν έχει καταβάλει, πιστεύω, μεγάλε προσπάθειε εκεί που είχε κάποια δυνατότητα επιρροή να εξασφαλίσει και τη συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα και οι στατιστικές δείχνουν ότι ακόμα δεν έχει επιτευχθεί αυτό σε ικανοποιητικό σημείο, αλλά υπάρχει ακόμα πολύ περιθώριο να επιτευχθεί αυτό και η Κομισιόν έπραξε πολύ και κυρίως είναι αποφασιστικό το ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα αξιολόγησης στι Βρυξέλλες πολύ πιο επωφελή και καλή από αυτή που έχουμε εδώ. Όταν λέμε για μια κουλτούρα αξιολόγηση, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πάντα να βλέπουμε σε ένα χρονικό ορίζοντα ο οποίος δεν περιορίζεται μονάχα στο τι γίνεται μισό χρόνο ή ένα χρόνο μετά το τέλος των ε, προγραμμάτων αυτών. Θέλουμε να δούμε ποιος ήταν ο αντίκτυπος σε ένα ορίζοντα πέντε ετών αργότερα. Ποιος είναι ο μακροχρόνιος λοιπόν αντίκτυπος αυτών των προγραμμάτων πλαισίου. Τελευταίο κομμάτι της παρουσίασής μου τι έχουμε μάθει από το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα και τι ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε στα πλαίσια του 8ου προγράμματος πλαισίου. Έχουμε δύο πυλώνες μέσα στην, στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και τεχνολογίας. Έχουμε καταρχήν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και μέσα σε αυτές είναι το να μπορέσουμε να έχουμε προγράμματα τα οποία έχουν σαφή στοχοθεσία, όπως παραδείγματος χάρη για την υγεία, για την ενέργεια και όλα Και τα λοιπά. Εδώ έχουμε μία εκ των άνω ε, προσέγγιση που λέμε ότι η Κομισιόν πρέπει να κάνει τα πράγματα αυτά μέσω του προγράμματος που δεν μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη από μόνα τους. Και φυσικά εδώ πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο η ποιότητα αυτών των προγραμμάτων, αλλά πρέπει να είναι και σχετικά με τις ανάγκες της ευρωπαϊκής κοινωνίας και βιομηχανίας. Από την άλλη πλευρά, ο άλλο πυλώνας είναι οι μεγάλες ιδέες. Είναι μεμονωμένα προγράμματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία σε ερευνητικό επίπεδο, έχουν σημασία για επενδυτές πολλές φορές. Εδώ χρειάζεται να τονίσουμε την αριστεία, την ποιότητα που θα είναι το κυριότερο κριτήριο. Και επίσης θέλω να τονίσω αυτά τα οποία στην επόμενη διαφάνεια τι είναι το σημαντικό για μας να προωθήσει η Κομισιόν. Καταρχήν θέματα τα προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την καινοτομία αλλά να έχουν και εφαρμογή, πρακτική εφαρμογή. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχάσουμε το βασικό στόχο που είναι να προωθήσουμε τις ε, βιομηχανικές εφαρμογές. Δεν πρέπει να περιοριστούμε μονάχα στα θέματα τα οποία αποτελούν ε, πρόκληση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα τα οποία είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαραίτητο να επιληθούν όπως είναι τα θέματα της δημόσιας υγείας, ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής όπου ανέφερα. Πρέπει επομένως να λάβουμε υπόψη την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για αυτά τα προγράμματα και τα οποία θα έχουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα μέσα στην ευρωπαϊκή, στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη χρήση εργαλείων τα οποία έχουν αποδείξει την αξία τους. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές αλλάζει συνέχεια τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Κομισιόν και ούτε οι επιστήμονες ούτε η βιομηχανία ξέρουν πού ακριβώς βρίσκονται. Έχουν τα ολοκληρωμένα προγράμματα, το NEST, τα μεμονωμένα προγράμματα θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν και κάποια σταθερότητα. Νομίζω ότι έχουμε μάθει πολλά από τα προηγούμενα προγράμματα πλαίσιο για το τι είναι καλό και το τι δεν είναι καλό και δεν χρειάζεται να αλλάζουμε συνέχεια το προστάσιο μας μέσα στα προγράμματα αυτά. Για τις μεγάλες ιδέες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το οδηγεί η καινοτομία και η έρευνα που περιλαμβάνει και κινδύνους ότι ίσως δεν θα είναι αποτελεσματικά αυτά τα προγράμματα. Είναι ο στόχος μας να προσελγίσουμε τους καλύτερους ερευνητές και τα καλύτερα ε, ιδρύματα στην Ευρώπη. Εδώ δεν έχει καμία σημασία η λεγόμενη δίκαια απόδοση, μονάχα η αριστεία. Και πιστεύουμε ότι εδώ οι μεγάλες προκλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από νέες καινούριε μεγάλες ιδέες οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα στο πρόγραμμα αυτό και το πιο σημαντικό επίση είναι το γεγονό ότι όλη αυτή η διαδικασία για την αντιμετώπιση των μεγάλων ιδεών και των σχεδίων να γίνεται με έναν τρόπο ο οποίο θα είναι διάφανο σε ό,τι αφορά την επιλογή και των ε, αξιολογητών και τη στρατηγική αξιολόγηση. Εν κατακλείδη, και πάλι, οι δύο μεγάλες προκλήσεις που αποτελούν το έργο της Κομισιόν θα πρέπει να καθορίσουν ποια είναι τα μεγάλα οι μεγάλες αυτές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Κομισιόν και αυτό δεν πρέπει να χάσει τον έλεγχο αυτής της, αυτού του ορισμού η Κομισιόν και να εξασφαλίσει ότι θα αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις με τα κατάλληλα όργανα. Και επίσης για τις ιδέες τόνισα προηγουμένως ότι τα μεμονωμένα προγράμματα και τα προγράμματα δικτύου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από μια δομή η οποία θα επιτρέπει όχι μονάχα μεμονωμένες ε, δράσεις από άτομα ή ιδρύματα, αλλά και αυξανόμενα προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν συνεργασία ερευνητών ή ιδρυμάτων. Ποιο είναι το όραμα λοιπόν της Ευρώπης που προκύπτει από όλα αυτά. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε αν ξεπεράσουμε την ιδέα της επικουρικότητας και της δίκαιας απόδοσης. Δεν περιοριστούμε λοιπόν σε αυτά σαν μόνο κριτήρια, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να κατανοήσουν ότι πρέπει να προωθήσει η Ευρώπη την ε, έρευνα και την ανάπτυξη. Επίσης, δεν θα πρέπει να περιοριστούμε σε ένα όραμα το οποίο αφορά μονάχα το εσωτερικό της Ευρώπης. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση παγκόσμιου ανταγωνισμού και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κατανοήσουν ότι τα προγράμματα πλαίσιο δεν είναι μια λεπτομέρεια, μια προστίκη σε σχέση με τα εθνικά ερευνητικά όργανα και προγράμματα, αλλά είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέμε τα εργαλεία τα οποία αλλάζουν και τη φύση του παιχνιδιού. Και επομένως δεν αρκεί να αλλάξουμε τεχνικά προγράμματα, πρέπει να υπάρξει ένα συντονισμός των εθνικών προγραμμάτων για να προχωρήσουν και γι' αυτό έχω προτείνει να υπάρξει και ένας πολλαπλασιασμός του προπολογισμού του προγράμματος πλαισίου κατά δύο ή τρεις φορές ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία προέρχονται από ευρωπαϊκές δράσεις έχουν αυτόματα μία προστιθέμενη αξία και αυτό ίσως θα μπορούσε να είναι και το σύνθημα του 8ου προγράμματος πλαισίου ότι μπορούμε να εδραιώσουμε την ευρωπαϊκή αριστεία έχοντας και μία όψη του γενικού πλαισίου του παγκόσμιου ανταγωνιστικού χώρου και συγχρόνως τονίζοντας την εσωτερική συνεργασία μέσα στην Ευρώπη. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ καθηγητά Ρίτσελ. Νομίζω ότι η παρουσίασή σας ήταν πολύ καλή, πολύ ακριβής, με πολλές πληροφορίες που μας δώσατε. Ε, ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσίαση, ε, γιατί την κατάλαβα και εγώ που δεν είμαι ειδικό. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, ε, όπως σας είπα, είδα ότι 9-10 άτομα ζήτησαν το λόγο, γι' αυτό θα σας ζητήσω να είστε σύντομοι. Ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό, διαφορετικά όμως δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ο κύριος Κορέα Δεκάμπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να συγχαρώ τον, κύριο, τον καθηγητή κύριο Ρίτσελ και την ομάδα του για την αξιολόγηση που έφεραν πέρα σε σχέση με το εκτό πρόγραμμα πλαίσιο και ως μέλος αυτού του κοινοβουλίου θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την μεγαλοψυχία, τη γενεοδορία αν θέλετε, που χρησιμοποίησε για να αξιολογήσει ένα πρόγραμμα που ξέρουμε όλοι ότι έχει πολλές ελλείψεις και κενά. Όπως και ο ίδιος όμως ε, έχει αναγνωρίσει, δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση έναντι του προγράμματος πλαίσιου. Έχουμε βέβαια το θέμα της ε, ανεπάρκειας των, των πόρων μόνο το 4% του συνδυασμένου προϋπολογισμού έρευνας των κρατών μελών αντιπροσώπευε το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο. Έχουμε επίσης το πολύπλοκο πρόβλημα του ότι εμείς δεν είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία με τους βιομηχανικούς κύκλους και ακριβώς όπως είπε και ο μιλτής ότι έχει μειωθεί η συνεργασία με τη βιομηχανία τα τελευταία χρόνια στα προγράμματα αυτά. Τα σχόλια τα οποία έχουν αναφερθεί σε σχέση με το πρόγραμμα πλαίσιο είναι συντριπτικά. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα αυτό γιατί εγώ θα είμαι μέλος αυτού του Επιστημονικού Συμβουλίου για την αρχή τουλάχιστον αυτής της θητείας και πιστεύω, του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Πιστεύω λοιπόν ότι μετά από όλα αυτά που έχουμε ακούσει πρέπει πράγματι να αλλάξει κάτι. Ο, ο μιλητής επίσης ανέφερε ότι υπάρχει έλλειψη ποιοτική πληροφορίας που κάνει πολύ δύσκολο να εξασφαλίσουμε αν παραδείγματος χάρη ο στόχος του 15% των κονδυλίων του έκτου προγράμματος πλαισίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν επετεύχθη ή όχι ένας τέτοιος στόχος. Αλλά είναι πεδαριώδες το να μην μπορούμε, το να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο, να ξέρουμε αν επιτεύχθη ή όχι ένας στόχος αυτού του είδους. Επίσης το θέμα της έλλειψης στρατηγικής, αυτά που, λέει, που είπε ο κύριος ο καθηγητής Ρίτσελ, μου φάνηκαν απόλυτα σωστά, γιατί δεν υπήρξε μια στρατηγική ενατένιση του έργου της έρευνας μέσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως αυτό μπορεί να οδηγεί και σε κατασπα... κατασπατάληση πόρων. Περαιτέρω, η... η αξιολόγηση, η γραφειοκρατία, το γεγονός ότι δεν περιμένουμε να τελειώσει ένα πρόγραμμα για να κάνουμε την αξιολόγησή του, αυτό οδηγεί πολλές φορές σε προβλήματα. Εγώ επίσης εγκαλούμε ιδιαίτερα από αυτή την ε, έκκληση που έγινε προς την Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Είπε ο κ. Ρίτσελ ότι και τα τρία θεσμικά όργανα είναι απαραίτητο να δράσουν για να τροποποιηθεί το πολύπλοκο σύστημα διαχείρισης και να το κάνουν πιο αποδοτικό. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, εγώ συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο καθηγητής Ρίτσελ, είναι θαυμάσιο το έγγραφο του καθηγητού για το μέλλον. Θέλω να σταθώ σε μερικά μονάχα παραδείγματα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ο πρόεδρος της ομάδας αξιολόγησης θεωρεί ακόμα ότι είναι δυνατό να διασωθεί το πρόγραμμα πλαίσιο 7, γιατί οι συστάσεις του ήταν θα πρέπει να προσπαθήσουμε τουλάχιστον το πρόγραμμα πλαίσιο 8 να έχει πιο απλούς κανόνες. Αλλά το ερώτημα είναι αν θεωρεί ότι είναι διασώσιμο μέσα σε εισαγωγικά και το πρόγραμμα πλαίσιο 7. Αυτό φυσικά δεν εμπίπτει στη δική σας εντολή, αλλά σίγουρα θα ήταν ενδιαφέρουσε οι πληροφορίε που θα μπορούσατε να μα δώσετε για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος και ζητώ συγγνώμη που κρατάω έτσι απειλητικά το σφυράκι του Προέδρου αλλά πραγματικά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι. Κύριε Νάμπερς, ευχαριστώ Πρόεδρε, κοιτάξτε, όταν έχουμε τόσο σοβαρά θέματα να συζητήσουμε, θα πρέπει να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Ρίτσελ για την παρουσίασή του και για τις προτάσεις που έκανε, που είναι αρκετά τολμηρές συμφωνούμε με τις προτάσεις αυτές πιστεύουμε ότι πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στους στόχους μας και η πρώτη άσκηση ας πούμε θα ήταν να αποφασίσουμε να μην κάνουμε κάποια πράγματα ε, διότι ε, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εστιάσουμε περισσότερο σε κάποια σοβαρά θέματα. Επίσης η εγκατάλειψη της αρχής της δικής απόδοσης, η δικής επιστροφής είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει σύμφωνος. Πιστεύω ότι εμείς τουλάχιστον πρέπει να το κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα από το Συμβούλιο. Τώρα για τους ελέγχους οι έλεγχοι κοστίζουν εάν όμως κοστίζουν ε, περισσότερο από ότι θα κόστιζε μια ενδεχόμενη απάτη τότε δεν πειράζει ας ε, έχουμε απλώς εμπιστοσύνη ας μην κάνουμε τους ελέγχους Εκείνο το οποίο είναι ιδιαίτερα τολμηρό είναι αυτό που ελέγχθη ότι θα πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες με τις ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες και πράγματι μόνο αν ανοίξουμε τις πόρτες μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε και καινοτομία. Επίσης από εκεί και πέρα για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή θα πρέπει να είμαστε λιγότερο περίπλοκοι στα δι... στις διοικητικές μας λειτουργίες αν θέλετε μετά για την ισότητα των δύο φίλων, βεβαίως Πράγματι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες αλλά όχι οπωσδήποτε ερευνήτριες αλλά επικεφαλής των ερευνητικών φορέων για να δείξουμε ποιο είναι το μήνυμά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την παρουσίασή σας και συμφωνούμε με τις περισσότερες προτάσεις σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ το ότι θα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, ναι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά εφόσον δεν έχουμε ε, πολύ χρόνο, τι να κάνουμε και υπάρχουν και μικρές καθυστερήσεις και κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσουμε, τελειώνουμε και τη συνέδριά μας. Τέλος πάντων θα προσπαθήσω να είμαι δίκαιος ο επόμενος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον καθηγητή Ρίτσελ για την παρουσίασή του και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι προ, προσπάθησε να ε, δει αν θέλετε τα πράγματα και μέσα στην προοπτική του 8ου πλαίσιου ε, προγράμματος πλαισίου. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις εδώ και 10 χρόνια με μέλος της Επιτροπής αυτής και ε, επί δέκα χρόνια νομίζω ότι συζητούμε περίπου τα ίδια πράγματα. Θυμάμαι πριν από την υιοθέτηση του 7ου προγράμματος ε, πλαισίου κάναμε μία λεπτομερή ανάλυση και είπαμε πόσο περίπλοκη είναι η διοίκηση, οι διοικητικοί κανόνες, οι διαδικασίες, οι εφαρμογές κτλ. Το ίδιο ε, λέγεται και στη χώρα μου, τη Γερμανία. Τα προβλήματα είναι γνωστά τελικά. Οπότε θα ήθελα ε, κάπου να ρωτήσω αφού και ενώπιση του 7ου προγράμματος πλαισίου είπαμε ότι πρέπει να διορθωθούν ορισμένα πράγματα τι έγινε τελικά. Υπήρξαν βελτιώσεις στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, πώς το δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, αλλά πώς το εκτιμάτε εσείς στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Τώρα όσον αφορά το άνοιγμα προς το εξωτερικό ε, και όσον αφορά κάποιες προσπάθειες που γίνονται για κάποιους εφαρμοστικούς φορείς που θα πάνε ε, θα μοιραστούν αν θέλετε Κοιτάξτε, γενικώ αυτοί οι φορεί δεν είναι και πολύ αγαπητοί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί ε, δυσκολεύουν με αυτή την έννοια και με τη διασπορά τέτοιων φορέων αν θέλετε δυσκολεύουν και οι έλεγχοι. Αλλά τι έχετε να πείτε για αυτούς τους εκτελεστικούς φορείς. Επίσης είπατε ότι ψάξατε και άλλες εναλλακτικέ δυνατότητες και τελικά δεν βρήκατε να υπάρχει μια εναλλακτική λύση οι καλύτερη από το πρόγραμμα πλαίσιο. Μιλήσατε για το ERC, μιλήσατε για υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες ε, όπου χρησιμοποιούνται χρήματα για έρευνα. Ε, δεν είμαι λοιπόν σίγουρη ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις καλύτερες, το ίδιο καλές όπως το πρόγραμμα πλαίσιο. Είπατε επίσης ότι ε, δεν θα πρέπει, θα να συμμετάσχει περισσότερο η βιομηχανία, δεν θα πρέπει να χάσει το ενδιαφέρον της για το πρόγραμμα πλαίσιο. Ωραία, σας ρωτώ εγώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τι γίνεται γιατί και στο 7ο ε, πρόγραμμα πλαίσιο είδαμε ότι και 25% μονάχα ε, των πόρων διατίθενται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν το πρόγραμμα πλαίσιο. Ευχαριστώ κύριο Τσουκαλάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον καθηγητή κύριο Ρίτσελ και την ομάδα του. Είναι κρίμα ότι το επόμενο θέμα μας δεν είναι η παρουσίαση της έκθεσης Μαριμών θα ακολουθηθεί το απόγευμα, θα μπορούσαμε με τη σύγκριση των δύο εκθέσεων να δούμε ότι συμπίπτουν στις ε, διαπιστώσεις, στις διαπιστώσεις που οδήγησαν στην αποτυχία της επίτευξης των στόχων της Λισαβόνας και νομίζω ότι είναι επίγον, επίγειο καιρός να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να εξακολουθήσω να μιλάω για τα red tape φαινόμενα των επιμέρους προγραμμάτων, όταν μου διαφεύγουν στην κεντρική πολιτική χάραξη οι στόχοι μιας ερευνητικής πολιτικής που θα μπορούσε να μας κάνει να πρωταγωνιστήσουμε σε αυτό που ο κύριος Μπαρόζο ονομάζει το όραμα του 2020. Δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη να αρχίζει να κομματιάζει τις δεκαετίες και το 2020 να αρχίσουμε να συζητάμε το όραμα του 2030 με ενδιαφέρει οι ευρωπαϊκές πατέντες να αρχίζουν να γίνονται πολυπληθέστερες από τις άλλες των ανταγωνιστών και με ενδιαφέρει να αναδεικνύονται τα κέντρα αριστείας στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Υπό την έννοια αυτή η έκθεση του καθηγητή κ. Ρίτσελ στο μότο που τελειώνει European Excellence through Global Cooperation and Competition θα έπρεπε ίσως να συμπεριλάβει και την ενδοευρωπαϊκή ανταγωνιστική διαδικασία, διότι τελικά αυτά τα ε, προγράμματα ε, αρχίζουν να μοιάζουν στις χρηματοδοτήσεις τους περισσότερο σαν επιδοτήσεις παρά σαν ανταγωνιστικά προγράμματα αρίστης έρευνας. Ε, ελπίζω ότι το απόγευμα, κύριε Πρόεδρε, στην παρουσίαση της εκθέσεως Μαριμών θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα γενικότερα διαρθρωτικά προβλήματα της ΕΡΑ και να συμπεριλάβουμε τα πάρα πολύ χρήσιμα και υπάρχοντα ήδη στην έκθεση Ρίτσελ αυτά τα γενικά συμπεράσματα τα απαραίτητα για τη διάκριση της ευρωπαϊκής έρευνας. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέω πρόεδρος. Ο κύριος Έλερ έχει το λόγο. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Ρίτσελ για την παρουσία του και για την παρουσίασή του και το γεγονός ότι αμφισβητεί και την αξία της συστηματικής των προγραμμάτων αυτών πλαισίου. Πιστεύω ότι πρέπει όλα αυτά να επηρεάσουν την ενδιάμεση αξιολόγηση των προγραμμάτων πλαισίου. Βλέπουμε πολλές φορές ότι δεν υπάρχει καμία συνέχεια, ότι δεν γίνεται καμία προσπάθεια όταν γίνεται η ενδιάμεση ε, ενδιάμεση αξιολόγηση των προγραμμάτων πώς θα επηρεαστούν τα προγράμματα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ήδη το έχουμε θέσει στα πλαίσια της αναθεώρησης του προγράμματος πλαισίου 7. Και θα θέλαμε να έχουμε και την άποψη της Κομισιόν ακριβώς για το πώς θα εκμεταλλευτεί αυτή την, ε, την, ε, την ενδιάμεση έκθεση, γιατί εμείς επιβάλλουμε μια ενδιάμεση έκθεση ακριβώς για να είναι υποχρεωμένη η Κομισιόν να εξετάσει την ε, επιτυχία του προγράμματος πλαισίου μέχρι εκείνο το σημείο. Μιλήσατε επίσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. <clears throat> Έχετε να δείτε πώς λειτουργεί αυτό με τα προγράμματα τα οποία εκτελούν διάφορες γενικές διευθύνσεις. Αυτά τα προγράμματα λοιπόν που είναι εκτός του προγράμματος αυτού και εκτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίες είναι αυτό που αναφέρατε, ότι ίσως θα πρέπει να έχουμε δομές οι οποίες, είναι, οι οποίες διαχειρίζονται από γενικές διευθύνσεις που είναι πιο κοντά στη βιομηχανία και ότι αυτό θα μπορούσε να κάνει μια διαφορά. <clears throat> Δεύτερον, ξεκινήσαμε με το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο μια σειρά από ανοίγματα προς την κατεύθυνση τρίτων χωρών και συνεργασία με τις τρίτες αυτές χώρες σε ποιο βαθμό αυτή η κίνηση προς τις τρίτες χώρες απεδείχθη εποφελής και το τελευταίο ερώτημα, όταν μιλάτε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εμείς πάντα μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις βάσει του ορισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φυσικά εξαρτάται από τον τομέα. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό το οποίο θεωρείται σαν μια μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με τον κλάδο και πολλές φορές έχουμε μεσαίες εταιρείες οι οποίες δεν είναι μικρομεσαίες σύμφωνα με τον αυστηρό ορισμό αλλά είναι η πηγή της καινοτομίας στους τομείς τους. Έχει νόημα λοιπόν κάτω οπότε τις συνδίκες να μιλάμε μονάχα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ κύριος Βάλσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αξιολόγηση του καθηγητή Ρίτσελ ήταν μεν λακωνική, αλλά ήταν και σαφέστατη στο ότι το πρόγραμμα αυτό δεν έχει καμία εναλλακτική λύση. Επομένω, τα προγράμματα πλαίσιο θα πρέπει να συνεχιστούν. Αλλά ο κύριος στόχος δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται, δηλαδή να υπάρξει μία προσέγγιση της βιομηχανίας με τους ερευνητές. Αυτό ενδιαφέρει και τις μεγάλες και τις μικρές εταιρείες, αλλά φαίνεται ότι όλο και λιγότερο υπάρχει αυτή η επαφή των επιστημόνων με τους ε, βιομηχανικούς κύκλους για τη θεραπεία των προβλημάτων, ο καθηγητή Ρίτσελ ανέφερε μερικέ προτάσει να μειώσουμε πραγματικά τη γραφειοκρατία. Και εδώ έρχομαι σε ένα σαφέ ερώτημα. Με ποιο τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε όταν γίνεται η αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων, των προγραμμάτων πλαισίου και συγκεκριμένα του 7ου προγράμματο πλαισίου, να επανέλθουμε στα ίδια ακριβώ ερωτήματα. Όπω αυτά που ακούσαμε τον καθηγητή Ρίτσελ σήμερα. Είναι απαραίτητο βέβαια για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα απορίσματα. Και το πραγματικό ερώτημα είναι πώς μπορούμε ήδη μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να επιφέρουμε όλες αυτές τις αλλαγές που αναφέρατε και που θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια πολιτική απόφαση προς την κατεύθυνση αυτή και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπατε εσείς ότι αυτές οι προτάσεις συγκεκριμένε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατό και όχι μονάχα μετά το τέλος ενός προγράμματος πλαισίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Ρίτσερς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς για αυτά που μας είπατε, αλλά να σας θέσω ένα ερώτημα για, τα, για το όραμα. Μία πρόκληση που αντιμετωπίζουμε για το μέλλον είναι να δημιουργήσουμε αυτόν τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνα, που είναι και ένα από του στόχου τη συνθήκη τη Λισαβόνας. Ανησυχώ ιδιαίτερα με τον περίπλοκο χαρακτήρα που χαρακτηρίζει κάποια από τα project, ε, παραδείγματο χάρη ότι θα πρέπει κάποια project να σέβονται το άρθρο 169 για να μπορούν να ενταχθούν σε αυτόν τον χώρο έρευνα. Α πούμε για την, για την Ελληνοσία. Τρία χρόνια χρειάστηκε να διαπραγματευτούμε ε, το project για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή. Στην βασική έρευνα συμφωνώ απόλυτα μαζί σα ε, ότι η το να ζητήσουμε ε, τα, από τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας είναι μια καλή λύση. Ανησυχώ όμως περισσότερο για την εφαρμοσμένη έρευνα και, την συμμετοχή τους, ε, και τη συμμετοχή των πανεπιστημίων, των εταιριών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν ξέρω εάν αυτό το εργαλείο θα είναι κατάλληλο για να μπορέσουμε να έχουμε πανευρωπαϊκά προγράμματα. Πιστεύετε ότι τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για κάποιες καινοτομίε ε, και τεχνολογικά ε, τεχνολογικές πρωτοβουλίες μπορούν να λειτουργήσουν. Έχετε άλλα πανευρωπαϊκά εργαλεία κατά νου για να μπορέσει, που, θα, θέλετε να εφαρμόσετε. Ευχαριστώ κυρία Ντεκαστήγιο. Ευχαριστώ καθηγητά Ρίτσελ, συγχαρητήρια. Πρέπει να σας πω ότι αυτή ήταν η καλύτερη παρουσίαση που έχουμε δει σε σχέση με την αξιολόγηση ενός προγράμματος πλαισίου, όχι μόνο σε ένα πολιτικό χώρο, αλλά πολλές φορές και σε ακαδημαϊκούς χώρους τους οποίους εγώ έχω συμμετάσχει στο παρελθόν. Και συγχαρητήρια για το τελικό σας σύνθημα με το οποίο συνοψίζεται την προσέγγιση του μέλλοντος, το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα πρόγραμμα πλαίσιο, το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο και επέκεινα του 8ου πρόγραμματος πλαίσιου. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει μια μεθοδολογία αξιολόγηση η οποία να έχει εφαρμοστεί με συνεχή τρόπο και επομένως να έχουμε κάποιους κανόνες εν καιρό, όπως έλεγε ο συνάδελφος μου ο κύριος Έλερ για το πώς να κάνουμε αυτές τις αξιολογήσεις. Έχουμε όμως μια σειρά από συμπεράσματα που ουσιαστικά έχουν επαναληφθεί στις τελευταίες αξιολογήσεις των προγραμμάτων πλαίσιο. Η έλλειψη συγκεκριμένα μια στρατηγικής ανατένισης για τα θέματα έρευνας, το θέμα της ύπαρξης μιας κουλτούρας αξιολόγησης, η επαναλαμβανόμενη αίτηση για διπλασιασμό ή τριπλασιασμό των κονδυλίων και τέλος η ύπαρξη μιας υπερβολικής διοικητικής πολυπλοκότητας. Από τα τέσσερα αυτά στοιχεία, το πιο δύσκολο για να αντιμετωπιστεί και το πιο επίμονο είναι για μένα το θέμα της διοικητικής πολυπλοκότητας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια γιατί αυτή τη στιγμή αποθαρρύνουμε όχι μόνο να τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και στο επίπεδο των ερευνητών που προχωρούν σε κατεύθυνση καινοτομίας, εμποδίζουμε να ευδοκιμήσουν προγράμματα τα οποία μπορεί να είναι καινοτόμα, αλλά δεν μπορούν να επιβιώσουν μέσα στη ζούγκλα του διοικητικού άχθους που χρειάζεται για να εγκριθεί ένα πρόγραμμα. Θεωρείτε τώρα εσείς ότι υπάρχει ένα σύνολο μέτρων τα οποία να είναι σωστά σχεδιασμένα ώστε μέσα στην προοπτική του 8ου προγράμματος πλαισίου να μπορέσουμε να έχουμε ένα δρόμο που θα μας οδηγήσει στην επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων που για μένα είναι τα πιο επίμονα, τα πιο δύσκολα για όλα τα προγράμματα πλαίσιο ή όχι. Ευχαριστώ. Κύριος Γκίρετ έχει το λόγο. Sam Προεδρεύεται μια ομάδα ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων και θα πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο κρίνονται κάποια project. Όταν έχουμε να κάνουμε τη δουλειά των εμπειρογνωμόνων, Διερωτώμε μήπως θα έπρεπε να ζητάμε και κάποια εξήγηση του γιατί ζητάμε τόσες πολλές διοικητικές διαδικασίες. Εάν δούμε πώς λειτουργήσαν τα προηγούμενα προγράμματα πλαίσιο, το έκτο ή το έβδομο, θα δούμε ότι υπήρχαν κάποια, ε, κάποια, κάποια στοιχεία τα οποία θα μας ε, οδηγήσουν σε κάποια συμπεράσματα και τα οποία θα είναι και χρήσιμα και εδώ. Διότι και εκεί υπήρχαν πολλοί εμπειρογνώμονες. Τώρα η ερώτησή μου. Στο έκτο πρόγραμμα πλαίσιο υπήρχε ένα Υπήρχε ένα συγκεκριμένο σχήμα το οποίο εφαρμόσατε και Επίσης, κύριε καθηγητά, μιλήσατε για τεράστια ποσά, για μεγαλεπίβολα προγράμματα. Μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα λύσεων τα οποία ε, πρότεινε το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ευχαριστώ πολύ καθηγητά Ρίτσελ για την παρουσίασή σας. Θα... Ε, η παρουσίαση ήταν ε, για το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο και δεν γίνεται αρκετός λόγος για το έβδομο. Ξέρω ότι δεν ήταν η δική σας δουλειά αυτό αλλά νομίζω ότι κάποια από τα προβλήματα που αναφέρατε είναι αντί να βελτιωθούν επιδεινώθηκαν στο 7 πρόγραμμα πλαίσιο αυτό ήταν το πρώτο μου σχόλιο και ένα δεύτερο είπατε ότι πρέπει να ε, αυξηθεί η συμμετοχή γυναικών ερευνητών. Ωραία, όμως για μένα το πρόβλημα δεν είναι τόσο οι γυναίκες, οι ερευνήτριες, αλλά οι νέοι ερευνητές εδώ στην Ευρώπη. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους να συμμετάσχουν. Γι' αυτό οι υποδομές μας θα πρέπει να είναι υποδομές που να τους βοηθούν βοηθούν τους νέους να μπορούν να συνδυάσουν τα οικογενειακά βάρη με την ε, ερευνητική δουλειά. Πρέπει λοιπόν πράγματι να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των νέων και των γυναικών. Είπατε επίση ότι πρέπει να προσελκύσουμε τους καλύτερους ερευνητές στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, ο στόχος μας ε, πρέπει να είναι πράγματι να έχουμε άριστους ερευνητές αλλά πρέπει να προωθήσουμε και την κινητικότητα εσείς είχατε επαφή με αυτούς τους άριστους ερευνητές τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε για να τους προσελκύσουμε να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευχαριστούμε πάρα πολύ ο καθηγητής Ρίτσελ τώρα θα πάρει το λόγο και θα προσπαθήσει να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις που ετέθησαν ίσως είναι ε, ε, πολλές οι ερωτήσεις αλλά πολλές ε, έμοιαζαν με προηγούμενες εν περιπτώσει ε, κύριε Ρίτσελ σας δίνω το λόγο και υποψιάζομαι ότι ε, μετά από την πολύ ενδιαφέρουσα συμμετοχή σας σήμερα ε, πολύ γρήγορα θα σας ξαναδούμε ναι με μεγάλη χαρά θα επανέλθω λέει ο κύριος Ρίτσελ θα ήθελα να απαντήσω και θα προσπαθήσω να ομοδοποιήσω κάπως τις ερωτήσεις ξεκινώ με την ερώτηση την προκλητική μπορεί να διασωθεί το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο η απάντηση είναι καταφατικά ναι διότι έγιναν πολλές βελτιώσεις σε πολλά σημεία του προγράμματος αυτού και ε, βεβαίως μπορεί να υπάρχουν και ορισμένα πράγματα που δεν διορθώθηκαν και θα διορθωθούν στο 8 ε, το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο είναι το πρόγραμμα πλαίσιο το οποίο έχει μια υγιεινή λογική όπου έχουν οριστεί στόχοι, υποστόχοι, υποστόχοι κτλ. μέχρι δηλαδή το επίπεδο των μεμονωμένων προγραμμάτων και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και πολύ καιρό και από για να μπορούμε όπως ελέγχθη ήδη να κάνουμε και τον έλεγχο μετά εκ των υστέρων και μια εκ των υστέρων αξιολόγηση. Δηλαδή το πρόγραμμα πλαίσιο έχει πάρα πολλές ευκαιρίες να πετύχει πάρα πολλές δυνατότητες και από εκεί και πέρα και πιστεύουμε ότι δεν θα είναι μόνο από επιστημονική άποψη επιτυχίας αλλά και από πολιτική άποψη. Τώρα για το διοικητικό φόρτο πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει η διοικητική, τη διοίκηση του ε, προγράμματος και αν δώστε εσείς το μήνυμα τότε πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσει και η Κομισιόν βεβαίω πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι διότι πρόκειται για τα χρήματα του φορολογούμενου από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να είμαστε να προσπαθήσουμε να μην κάνουμε πολύ λεπτομερείς ελέγχους ή ε, δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό που γίνεται μέχρι τώρα και το οποίο ουσιαστικά ε, αποθαρρύνει τους ερευνητές να ζητήσουν ευρωπαϊκά χρήματα για την έρευνά τους. Αν αποθαρρύνουμε λοιπόν τους ερευνητές ουσιαστικά ε, βάζουμε τρικλοποδιά ε, στον ανταγωνισμό και στη βελτίωση του ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει κάπου να δώσουμε το μήνυμα ότι έχουμε, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένο στο θέμα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία για τους ελέγχους τώρα για τις τρίτες χώρες και τη συμμετοχή τους το αναφέραμε το θέμα αυτό και υπάρχουν ε, πολύ καλές επαφές με αναπτυσσόμενους χώρους με την Ινδία, με τη Βραζιλία και διαπιστώσαμε ότι ε, ε υπήρχαν προβλήματα στο παρελθόν ναι, το μεγαλύτερο η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο με τους περισσότερους ερευνητές και επιστήμονες είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής. Στο έτο πρόγραμμα πλαίσιο δώσαμε μόνο 2 εκατομμύρια ευρώ για τη συνεργασία αυτή. Άρα πιστεύουμε ότι ναι μεν ε, έχουμε μια κάποια συνεργασία αλλά με αλλά πρέπει να ενισχυθεί σαφώς. Επίσης θα ήθελα να σας πω, να σας δώσω ένα παράδειγμα το που χρησιμοποιήθηκαν εξαιρετικά οι πόροι και το παράδειγμα αυτό είναι η ευρατόμο. Ε, πραγματικά είναι παραδειγματικός ο τρόπος οργάνωσης ε, ορισμού των προγραμμάτων, σχεδιασμού των προγραμμάτων της Ευρατόμ. Αν μπορούσαμε να μιμηθούμε ή να πάρουμε σαν υπόδειγμα την Ευρατόμ, νομίζω ότι θα κάναμε πολλά καλά πράγματα στην Ευρώπη. Κάτι άλλο τώρα, στόχος ήταν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 14% το αυτό να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Δεν το επιτύχαμε το στόχο αυτό. Ίσως λοιπόν πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική άγουσα. Ίσως θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αντίθεση με τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων. Ε, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, όντως μεγάλες επιχειρήσεις δεν έχουν πρόβλημα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν πρόβλημα θα πρέπει να δούμε ότι ε, κάποιες μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πολύ ε, ε, είχαν συγκεκριμένο επιστημονικό πρόβλημα αν θέλετε για το οποίο επιζητούσαν λύση ε, μπόρεσαν να ε, συμμετάσχουν αλλά γενικότερα το πρόβλημα μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπάρχει τώρα όσον αφορά την μη διάκριση και την ισότητα των φύλων βεβαίως και βεβαίως πρέπει να προσέξουμε τους νέους αντίθετα με αυτό που πιστεύει ο περισσότερος κόσμος. Οι νέοι άνθρωποι δεν ε, έχουν πρόβλημα λόγω ε, μισθού αν θέλετε. Έχουν πρόβλημα γιατί έχουν άλλα προβλήματα. Πρώτα πρώτα λοιπόν πρέπει να ε, φροντίσουμε να έχουμε καλή συνεργασία και εκτός Ευρώπης, Ιαπωνία κτλ. Δεύτερο, καλές υποδομές και τρίτο, να δούμε ότι να φροντίσουμε τα πανεπιστήμια να είναι καλά, να κάνουν καλή έρευνα που μπορούν να συμμετάσχουν και να έχουν, δίνουν τη δυνατότητα για, για σταδιοδρομίες στους νέους. Ε, νομίζω να, προχτές ήμουνα με τον Ιάπωνα πρέσβη στο Βερολίνο και είδαμε ότι όλο και λιγότεροι Ιαπωνέζοι έρχονται στην Ευρώπη. Στην, στο Βερολίνο ε, η γλώσσα είναι σημαντικό πρόβλημα ε. Ε, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Νομίζω ότι Απ' την άλλη μεριά δεν χρειάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ασχοληθούμε με την ανταγωνιστικότητα. Τα κράτη-μέλη ασχολούνται επαρκώς με αυτό. Εμείς εκείνο που πρέπει να φροντίσουμε είναι να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών, μια άμυλα μεταξύ των κρατών μελών για να μπορέσουμε να ε, γίνουμε αρκετά καλοί για να ε, ε, ενισχυθούμε σε σχέση με την Ιαπωνία, την Κορέα, τις Ηνωμένε Πολιτείε. Σας ευχαριστώ πολύ καθηγητά Ρίτσελ για την παρουσίασή σας και για τις απαντήσεις σας αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο να μπορούμε να πούμε ότι ήσασταν πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμος στην αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Νομίζω ότι έχετε ακούσει αγαπητοί συνάδελφοι την παρουσίαση των προβλημάτων. Τώρα, η διαδικασία που προβλέπετε βέβαια δεν είναι ακόμα σαφής. Τόνισε ο καθηγητής Ρίτσελ ότι εξαρτάται από τα μεγάλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Εγώ προτείνω Ακολουθώντα αυτό που ζήτησε ο καθηγητής Ρίτσερ, να δημιουργήσουμε μια ομάδα εργασίας που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό και να προσπαθήσουμε με αυτή την ε, άτυπη ομάδα εργασία να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Η επίσημη συζήτηση βέβαια θα γίνει στη συνέχεια. Να φτιάξουμε μια άτυπη ομάδα εργασία η οποία δεν θα έχει βέβαια δεσμευτικό χαρακτήρα τα πορίσματά τη, αλλά αυτό θα μα επιτρέψει να προχωρήσουμε σε μια ταχύτερη συζήτηση. Φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνείτε και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Ας το αποφασίσουμε λοιπόν αυτό. <clears throat> Θα ήθελα να σας παρακαλέσω λοιπόν κάθε πολιτική ομάδα να μας κάνει μια πρόταση για ένα εκπρόσωπο και να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο για να επιταχύνουμε λιγάκι τα πράγματα. Βλέπετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που αρχίζει να γίνεται κουραστική. Θέλω να σα ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ. Μα βοηθήσατε πάρα πολύ, όχι μόνο πνευματικά, αλλά μα κάνετε και προτάσει για να μπορέσουμε να βρούμε ένα νέο δρόμο. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ähm, Κυρίες και κύριοι, <clears throat> συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Ερχόμαστε στο σημείο 5, 4 μάλλον. Πρόκειται για τα μέσα τα οποία εφαρμόζονται στο σχέδιο ανάκαμψης για τα θέματα ενέργειας. Έχουμε μισή ώρα γιατί ο κύριος Επίτροπος θα πρέπει να πάει σε μια άλλη συνεδρίαση. Θα ακούσουμε τις απόψει του και θα μπορέσουμε ίσως να θέσουμε μερικά ερωτήματα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλήρη συζήτηση. Με μεγάλη χαρά λοιπόν θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Επίτροπο Πίμπαλκ, που είναι φυσικά η τελευταία του παρουσία στην Επιτροπή μας <clears throat> ως αρμόδιος για τα θέματα ενεργείας είχαμε μεγάλη χαρά που μπορέσαμε να συνεργαστούμε μαζί σας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας. Όταν αλλάζει χαρτοφυλάκιο ένας επίτροπος, είναι από μία πλευρά κρίμα που δεν είσαστε πια παρόν, παρά το γεγονός ότι είναι πολλές φορές πολύ ικανός και ο αντικαταστάτης σας. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάντως για τα πέντε χρόνια εξαιρετικής συνεργασίας μαζί σας. Σας δίνω το λόγο. Uh, ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους σας γιατί πραγματικά ήταν ε, μια μεγάλη ευχαρίστηση για μένα να συνεργαστώ μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια. Και σήμερα ήθελα να μιλήσω στην Επιτροπή σας ε, για, μια, για την πρόοδο που είναι πολύ θετική για την εφαρμογή του, σταδίου, του, του προγράμματος εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας. Ήδη έχουμε το πόσο σημαντικά είναι τα, ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανάκαμψη ε, της ε, οικονομίας και για την ε, ενεργειακή προμήθεια φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ούτως ή άλλως, κυρίως όσον αφορά το, τα project που αφορούν τα σημεία διασύνδεσης για το φυσικό αέριο και, την, και και τον ηλεκτρισμό, όπως επίσης ε, και τα σχέδια για την ε, δέσμευση και την αποθήκευση άνθρακα, είναι project τα οποία είναι ε, ουσιαστικά για την, για την Ευρώπη. Τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ε, δοθεί για τα διάφορα ενεργειακά project. Ε, μετά την, ε, μετά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη, το οποίο υποβάλαμε τον Νοέμβριο του 2008 ένα συμβου... και που επιβεβαιώθηκε από το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, η Κομισιό είχε δεσμευτεί να υποβάλει μια, ένα κατάλογο συγκεκριμένων project. Εμείς απαντήσαμε άμεσα και ε, τον Γενάρη του 2009 προτείναμε και τον συγκεκριμένο κανονισμό. Ε, χάρη στις ε, επικοδομητικές συζητήσεις ανάμεσα στα κοινοτικά θεσμικά όργανα καταλήξαμε σε μια συμφωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία υλοποιήθηκε τον πέρυσι τον Μάιο. Στην συνεδρίαση της συνδιαλλαγής που έγινε στις 18 Νοεμβρίου επιτρέψαμε την υιοθέτηση και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας για το 2009, 2010. Συγγνώμη. Πρέπει να πούμε όμως ότι αυτό το σχέδιο δεν ξεκίνησε από το μηδέν. Είχαμε και κάποια προηγούμενα βήματα τα οποία είχαν γίνει. Ο κανονισμός για το EP επιτρέπει να, του Ευρωπαϊκού Σχέδιου δηλαδή, επιτρέπει να εφαρμόσουμε κάποιους συγκεκριμένους στόχους, να υπάρχει ανάκαμψη της οικονομίας, να προσφέρουμε δυνατότητες για συμπληρωματικές θέσεις απασχόλησης και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και κατά τη διάρκεια της φάσης συνεργασίας. Όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, διευκολύνουμε την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ε, εσωτερικής αγοράς Δημιουργώντα δημιουργώντας και συμπληρώνοντας τις, τους κρίκους της αλυσίδας που λείπουν. Δείχνουμε αλληλεγγύη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης ε, μετά την κρίση του χειμώνα του 2009 και επιταχύνουμε και την υλοποίηση των στόχων του 2020 εφαρμόζοντας στρατηγικές και τεχνολογίες με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα. Ε, ήθελα να πω επίσης ότι πρέπει να διευκολύνουμε και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό και να στεφθεί με επιτυχία. Τους τελευταίους μήνες εργαστήκαμε σκληρά έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου ε, έχει τεθεί σε τροχιά. Λίγες μέρες μετά την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο για το πρόγραμμα αυτό ε, σε αρχές του Μαΐου έγινε η προκήρυξη του διαγωνισμού που καλύπτει τους τρεις τομείς και το σύνολο του του προϋπολογισμού. Η τελική ημερομηνία ήταν 15 ε, Ιουλίου του 2009. Κατά τη διάρκεια της ε, περίοδου αυτής ε, υποστηρίξαμε όλα, όλους τους φορείς πρόθεσης των ενδυνάμει project οργανώνοντας ενημερωτικές συναντήσεις και ενημερώνοντας το website του Ευρωπαϊκού Σχεδίου απαντώντας σε ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος. Έτσι όπως περιμέναμε ούτως ή άλλως, ο διαγωνισμός αυτός είχε πολύ θετικές ε, ε, απαντήσεις από πλευράς της βιομηχανίας. 87 ε, απαντήσεις υποβλήθηκαν, 46 για τα σημεία για τα σημεία διασύνδεση, 29 για, τις υπεράκτιες, ε, για τα υπεράκτια αεολικά πάρκα και 12 για, τις, για τα project ε, δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. Όλε οι προτάσει αυτέ που υποβλήθηκαν ήταν πάρα πολύ καλέ και σεβόντουσαν τα κριτήρια τα οποία ε, συμπεριλάμβανε ο κανονισμό συμμορφωνόντουσαν επίση και το εξετάσαμε και κατά πόσο συμμορφωνόντουσαν και με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υπήρχαν συγκεκριμένου και συγκεκριμένα σημεία τα οποία ήταν κοινά σε όλα αυτά τα project και τα οποία τα λάβαμε υπόψη μα όταν τα αξιολογούσαμε. Παραδείγματο χάρη η ορίμανση του σχεδίου, η οριμότητα μάλλον, κατά πόσον δηλαδή η εφαρμογή αυτού του project θα μπορούσε να συνεισφέρει βράχη πρόθεσμα στην οικονομική ανάκαμψη Δεύτερον, ε, κατά πόσον, τι, τι βοήθεια, τι κοινοτική βοήθεια χρειαζόταν για την ε, εφαρμογή του project αυτού και κατά πόσον τα project αυτά συνεισέφεραν στους ευρύτερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπρεπε να τονίσουμε και πρέπει να τονίσουμε επίσης ε, την συνεισφορά των κρατών μελών στην έγκαιρη εφαρμογή του project, παραδείγματο χάρη επιταχύνοντας τις διαδικασίες για την έκδοση εγκρίσεων ή αδειών. Δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να συμμορφώνομαστε με τους κανόνες ανταγωνισμού και τις, γενικότερα τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ε, για την ε, ενέργεια. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε διαφανείς ε, και κανόνες που δεν εισάγουν διακριτικές αντιμετωπίσεις και στον τομέα της, του, ηλεκτρονισμού, του ηλεκτρισμού του φυσικού αερίου. Αυτό είναι απαραίτητο έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να υποφεληθεί πλήρως από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Άγραψη της Οικονομίας. Η αξιολόγηση των προτάσεων για, την, για τα αιωλικά, για τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα και την για τα project δέσμευσης ε, άνθρακα έχει ολοκληρωθεί. Στις 16 Οκτωβρίου ε, η Επιτροπή ε, ολοκλήρωσε την μελέτη και την έγκριση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε σε όλη την διαδικασία της επιτροπολογίας και για τα παράκτια, υπεράκτια αιωλικά πάρκα και για το, τα project δέσμευση του, του άνθρακα θα ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία και θα τεθούν σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του χρόνου. Η αξιολόγηση τώρα της διαδικασίας για, τα, για τους σημεία διασύνδεσης κράτησε λίγο παραπάνω λόγω ακριβώς του μεγάλου αριθμού των project που είχαν υποβληθεί και λόγω ακριβώς και της περιπλοκότητας των project αυτό για τα σημεία διασύνδεσης. Θα υποβληθούν ε, στην, αξιο, στην Επιτροπή Αξιολόγησης στις 18 Δεκεμβρίου ε, η, μελέτη, η εξέταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα γίνει μετά, μετά τις 18 Δεκεμβρίου. Ε, θα υιοθετηθεί η απόφαση της Κομισιόν, περιμένουμε, τον Φεβάριο του 2010. Όπως ξέρετε, ο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ανάκαμψη ε, προβλέπει ότι θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2010 η Κομισιόν να έχει δεσμεύσει συγκεκριμένα κονδύλια. Το σχέδιό μας είναι να δεσμεύσουμε το σύνολο του προϋπολογισμού 3,86 ε, δισεκατομμύρια ευρώ από το σύνολο των 3,98 δισεκατομμυρίων ευρώ και όλα αυτά μέχρι την άνοιξη του 2010 για να έχουμε τα μεγαλύτερα κίνητρα αν θέλετε τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Η βιομηχανία ε, ε, απήντησε άμεσα ακριβώς ο λόγο το ότι επιλέξαμε τα συγκεκριμένα και τα καλύτερα project και γιατί ζητήσαμε ακριβώ την βοήθεια. Το Παγκόσμιο μειώσει, μας ζήτησε ούτως ή άλλως να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους ε, προγράμματα ε, κινήτρων. Και το ευρωπαϊκό, σχεδίο, δηλαδή, το ευρωπαϊκό σχέδιο δηλαδή πιστεύω ότι ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Και ε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό γιατί η Κομισιό ε, μπόρεσε να εφαρμόσει ένα τέτοιο τεράστιο πρόγραμμα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου. Τώρα, πέραν της, ε, παρα, της παρουσίασής μου σήμερα θα πρέπει να σας πω ότι στο επόμενο Συμβούλιο Ενέργειας στις 7 ε, Δεκεμβρίου θα συζητηθεί το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ανάκαμψη της Οικονομίας και το Μάρτιο του 2010 η Κομισιό θα υποβάλει ε, ε, θα υποβάλει μια έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 88 του κανονισμού και, και τότε θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού αλλά και όσον αφορά του κινδύνους εφαρμογής των διαφόρων project. Κατά την άποψή μου το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης της Οικονομίας πιστεύω ότι μπορεί να δώσει μια άμεση έγκαιρη και αποτελεσματική απάντηση στην σημερινή κρίση. Το σχέδιο αυτό είναι το απαραίτητο εργαλείο έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η εφαρμογή των διαφόρων ε, διαρθρωτικών ε, project ε, δεν θα καθυστερήσει και απαντά στις ανάγκες του... Του... ευρωπαϊκού κλάδου και της ενέργειας. Και όλα αυτά βέβαια θα, θα εξαρτηθούν από την επιτυχημένη εφαρμογή των project. Και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και το... τα θεσμικά όργανα της κοινότητας και οι... τα κράτη-μέλη και οι διάφοροι επιχειρηματίες που συμμετέχουν πρέπει να κάνουν το ό,τι μπορούν καλύτερο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Άκρη Ψυχονής είναι συγκυριακό πρόγραμμα το οποίο ε, οφείλεται στην κρίση λύση. Όμως θα πρέπει να συνδέεται και με τις άλλε πρωτοβουλίε που αναλαμβάνονται στον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο και για τα διαρθρωτικά ενεργειακά προγράμματα και για τα επόμενα χρόνια. Και επίσης θα πρέπει να βοηθήσει και την ενεργειακή ασφάλεια. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Εξυπτά ζήτησαν ήδη το λόγο. Θα ξαναπώ αυτό που είπα πριν, να είμαστε όλοι σύντομοι για να μπορέσουμε να τελειώσουμε έγκαιρα, γιατί ο κύριος Πίπαλξ πρέπει να πάει και σε μια άλλη συνεδρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε για την ε, συνεργασία τα τελευταία χρόνια. Έχω δύο ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα ανάκαμψης της οικονομίας. Χάρηκα ιδιαίτερα που τα καινούργια κίνητρα ε, συζητήθηκαν και ε, αποφασίστηκαν. Ωστόσο δεν χάρηκα ιδιαίτερα για το γεγονός ότι δεν προβλέπεται στήριξη για τις υποδομές σε ορισμένες χώρες που τις χρειάζονται κεντρική Ανατολική Ευρώπη παραδείγματος χάρη γιατί το Βέλγιο υποστηρίζεται ενώ έχει ήδη κάποιες βασικές ε, βασικά interconnector το Βέλγιο παραδείγμα ε, ε, ενώ άλλες χώρες που δεν έχουν ήδη κάποιες υποδομέ δεν μπορούν να στηριχθούν λόγω όλων αυτών θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα πρόεδρε πρώτον βλέπετε να μπορεί να ε, δοθεί ε, περισσότερη χρηματοδότηση στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη δεύτερον ε, μέσα στο ε, επικείμενο σχέδιο δράσης για την ενέργεια θα περιλαμβάνονται και στοιχεία για τη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς κύριε Επίτροπε. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ευχαριστώ για όλα αυτά που έχετε πράξει μέχρι τώρα. Μήπως μπορείτε να συνεχίσετε να πράτετε τόσα θετικά πράγματα για μας και στο μέλλον. Έχετε μεγάλη εμπειρία στα θέματα της ενέργειας και γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω το εξής. Να απαντήσετε ποια είναι η σύσταση που θα διαβιβάσετε στον διάδοχό σας για την εφαρμογή περαιτέρω ενεργειών στον τομέα της ενέργειας ποιες μεθόδους εργασίας επίσης θα προτείνετε στον διάδοχό σας να υιοθετήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σφόμποντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Και εγώ θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στο έργο σας και στην πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με, με εσάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως στην Επιτροπή Ενέργειας και Έρευνας για το θέμα του σχεδίου ανάκαμψης. Χαίρομαι που πάρα πολλά κονδύλια μπορούν να αποδοθούν ήδη την άνοιξη αφού φτάσουμε στον τελικό γύρο διαπραγματεύσεων. Αυτό ήταν κάτι το οποίο εμείς το απαιτήσαμε γιατί αυτό το νόημα έχει και ένα πρόγραμμα ανάκαμψης. Έπρεπε να τρέξω στην ακρόαση μέσα σε εισαγωγικά της κυρίας Άστον. Τρέχω πάνω κάτω, αλλά ήθελα να αναφερθώ στο ερώτημα που έθεσε η, η Ουγγαρέζα συνάδελφός μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την ασφάλεια σε ό,τι αφορά την ασφάλεια τροφοδοσίας με φυσικό αέριο που θα αναφερθεί σε αυτήν και ο κύριος Φιδάλ Κουάδρα στην έκθεσή του αργότερα. Είναι απαραίτητο στο βαθμό του δυνατού τα κονδύλια να δαπανηθούν τώρα και στα επόμενα χρόνια για τη βελτίωση των διασυνδέσεων, ιδίως στις υποδομέ φυσικού αερίου, γιατί υπάρχει το παράπονο ότι αυτό που προτείνετε εσεί μέσα σε τρία χρόνια να περατωθεί αυτή η υποδομή, ότι είναι ανεπαρκής ο χρόνος που είναι στη διάθεσή μας. Θέλω να χρησιμοποιηθεί όλος ο χρόνος που είναι απαραίτητος, αλλά όλα αυτά να βασίζονται σε στερεές, σε στα, σταθερές οικονομικές προβλέψεις. Εγώ θα ήθελα λοιπόν το πρόγραμμα ανάκαμψης να συμβάλλει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στις χώρες που υπάρχει και η μεγαλύτερη ανάγκη για υποδομές ενέργειας να εξασφαλίσει αυτές τις ε, υποδομές και επομένω και την ασφάλεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο και γενικά σε ενεργειακούς πόρους. Επομένως το θέμα των διασυνδέσεων για, για την ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να έχουμε πληροφορίε που θα μα βοηθήσουν να προχωρήσουμε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τον κανονισμό για την ασφάλεια τροφοδοσία ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ποδηματά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη σύντομη παρουσίασή του και για την παρουσία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ και νομίζω ότι εκφράζω το σύνολο των συναδέλφων εδώ ότι ο Επίτροπος Πίμπαλξ έδωσε στο χαρτοφυλάκιο της ενέργειας υπόσταση, το αναβάθμισε θεαματικά και συνέβαλε ώστε να καταστεί ένα από τα πιο περιζήτητα χαρτοφυλάκια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εκφράσω την ευχή ο διάδοχός του στο χαρτοφυλάκιο της ενέργειας να συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση και με την ίδια επικοδομητική διάθεση. Σε ό,τι αφορά την, το σχέδιο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας και τις επισημάνσεις που κάνατε, ε, ήθελα να θέσω ορισμένα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα αναφερθήκατε στα κριτήρια της οριμότητας ενός έργου, στην ορίμανση ενός έργου, σε ένα από τα βασικά κριτήρια για την ένταξή του στα επιλέξιμα έργα και ήθελα να επιμείνω λίγο ε, σε αυτό το σημείο κατά πόσο δηλαδή η οριμότητα ενός έργου είναι και θα παραμείνει μέχρι τη διαμόρφωση του τελικού καταλόγου των επιλέξιμων έργων καθοριστικό στοιχείο και να συνδυάσω αυτό το ερώτημα με το γεγονός ότι το, το 1 τέταρτο κύριε επίτροπε όπως γνωρίζετε ε, του ποσού των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ποσό ενός δισεκατομμυρίου ε, ευρώ έχει αποφασιστεί να κατευθυνθεί προς τα έργα συλλογής και αποθήκευσης άνθρακα έργα τα οποία είναι γνωστό ότι ακόμη βρίσκονται στο στάδιο ε, της έρευνας. Το δεύτερο σημείο, σε συνέχεια και της παρέμβασης του συναδέλφου Χάνες Βόμποντα αφορά στα ιδιαίτερα προβλήματα ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης και να επιμείνω λίγο για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που αντιμετώπισε και σοβαρά προβλήματα ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού κατά τη διάρκεια της ε, περσινής ρώσο ουκρανικής κρίσης και για την οποία οι διασυνδέσεις φυσικού αερίου παίζουν καθοριστικό ρόλο είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. υπάρχουν λοιπόν στον αρχικό κατάλογο των επιλέξιμων έργων ε, ορισμένα έργα που αφορούν ειδικά βελτιώνουν αισθητά την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού σε αυτή την περιοχή και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στον, ε, στον itgi και στον, ε, και στον igb. ειδικά σε ό,τι αφορά τον, τον τον ITGI ε, εδώ και αρκετά χρόνια έχει χαρακτηριστεί έργο μεγάλου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Η κατασκευή του έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά και υπάρχει ένα τμήμα του το οποίο ήδη λειτουργεί. Ε, ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, με δεδομένο ότι είναι ένα από τα πιο ώριμα έργα, είναι ένα από τα πιο προχωρημένα έργα προς την κατεύθυνση ε, ενός από τους κεντρικούς στόχους που έχουμε θέσει στο ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών, ε, κατά πόσο η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει πολιτικά ε, την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τον Επίτροπο τον κύριο Πίμπαλξ για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία σε όποιον τομέα επιλέξει ε, και στο μέλλον και να έχει την ίδια επιτυχία όπως και τώρα. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω... Ε, ότι για τα ε, project δέσμευση συλλογή και αποθήκευση άνθρακα. Ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκα τα, τα project αυτά και θα ήθελα να ξέρω έχουν συναυθεί συμβόλαια, έχουν υπογραφεί συμβόλαια, έχουν γίνει συμβάσει ε, και λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα της τεχνολογίας θα μπορέσετε να εφαρμόσετε όλο τον προϋπολογισμό που προβλέπετε για το 2009-2010. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ σύντομα όλα αυτά που είπατε και πολύ καθαρά. Κύριος Χατζημαρχάκης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όχι μονάχα γιατί ήσασταν τόσο συχνά εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά ήσασταν και αυτός ο οποίος εξε... επεζήτησε να έχει επαφές και με τους βουλευτές και γι' αυτό θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Και όπως είπε και η κυρία ε, Ποδηματά, έχετε πράγματι ε, αντιμετωπίσει με μεγάλη επιτυχία το χαρτοφυλάκιό σας. Νομίζω ότι έχετε αντιμετωπίσει επίσης σωστά το θέμα των ανανεωσίμων ενεργειών με το οποίο ε, ασχολήθηκα και εγώ και δείξατε μεγάλη επιτυχία στο θέμα της αιωλικής ενέργειας. Αυτό είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και αυτό το οποίο θα ήθελα να εξασφαλίσω είναι ότι όλα αυτά τα προγράμματα να μπορέσουν να εφαρμοστούν, να έχουμε μια ανταγωνιστικότητα στον παγκόσμιο χώρο, να είμαστε ανταγωνιστικοί γιατί έχουμε μεγάλη ισχύ σε ό,τι αφορά τα αιωλικά πάρκα και την αιωλική ενέργεια. Αλλά έχουμε όλο και προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Οι ρότορες γίνονται όλο και πιο μεγάλοι, πιο ε, δύσκολο είναι να μεταφερθούν και να εγκατασταθούν αυτοί οι ρότορες των ανεμογενετριών. Θα ήθελα να συνδέσω αυτό το οποίο συζητούμε τώρα με τα θέματα που μας, που μας απασχόλησαν το πρωί περισσότερο, τα θέματα της έρευνας. Μήπως θα μπορούσε να υπάρχει πιο έντονη σύνδεση με προγράμματα έρευνας όπως το 7ο και το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά και θέματα συνεργασίας με φορείς όπως οι χαλιβουργίες που κάνουν έρευνα στον τομέα αυτό της αντοχής των υλικών που έχει σχέση με τις ε, ανεμογεννητρίες. Ξέρω ότι εσείς αλλάζετε τώρα χαρτοφυλάκιο Ξέρουμε ότι για κάποιες αρμοδιότητες από το τωρινό σας χαρτοφυλάκιο θα περάσουμε στην Επίτροπο που είναι αρμόδια για τα θέματα ε, κλίματος, κλιματικής αλλαγής. Επίσης κάποια θα πάνε στην εσωτερική αγορά και στην διεύνηση. Το ερώτημά μου είναι κατά πόσο θα μπορέσει ο διάδοχός σας να είναι τόσο αποτελεσματικός όσο εσείς που είχατε ένα πληρέστερο χαρτοφυλάκιο. Ο κύριος Όντι έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ με τους συναδέλφους ε, τον Επιτροπό για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση, μία συγκεκριμένη ερώτηση. Έχουμε εμπιστοσύνη, έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη σε εσά. Και ήθελα να ρωτήσω, ειλικρινά δεν πιστεύετε ότι αυτή η θετική ορολογία που χρησιμοποιείτε, το λεξιλόγιο, το θετικό, ότι όλα πάνε καλά, όλα προχωράνε κτλ. Δεν είναι ότι είναι λάθος, αλλά υπάρχει ένα ρήγμα ανάμεσα στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση και τους, πολίτες. Ε, αυτό το ρήγμα και αυτή η ρήξη δεν προέρχεται ε, από, την, το ότι δεν ότι δεν έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, ε, τουλάχιστον στα μάτια των, των πολιτών από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενέργεια δεν, έχει, δεν ήταν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Όμως λέγαμε συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει εκείνο, θα κάνει το άλλο, θα κάνει το άλλο για την, για την ενέργεια. Ε, τώρα βέβαια με τη συνθήκη της Λισαβόνας διευρύνονται οι, οι αρμοδιότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά την ε, ασφάλεια ανεφοδιασμού. Όμως υπάρχουν στοιχεία για τα οποία δεν είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματο χάρη εμάς, τα πυρηνικά μας κέντρα ας πούμε, πα, παραγωγής ηλεκτρισμού χαλάνε δεν φταίει σε τίποτα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σημείο αυτό. Και ρωτώ, ε, μήπως για, για, τις, για, τα, για τις διαρθρώσεις, για τις υποδομές, μήπως... Ε, εδώ είμαστε μάρτυρες ε, μιας ε, αποτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάζουμε χιλιάδες δισεκατομμύρια ευρώ στο τραπέζι. Ε, και, ρωτώ έχουμε κάνει αρκετά όμως πράγματα, γιατί λόγω των προκλήσεων δεν μπορούμε να λέμε ιστορίες στους πολίτες, διότι αλλιώς οι πολίτες δεν πρόκειται να μας πιστέψουν. Ε, οι, οι προεκλογικές εκστρατείες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν μπορούμε να λέμε ψέματα συνέχεια. Έχω άλλους τρεις ομιλητές και κλείνω τον κατάλογο αγοριτών γιατί δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε τον κύριο Επίτροπο Περιτέρο. Ο κύριος είναι επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Επίτροπε, εγώ θα ήθελα να προσθέσω και τις δικές μου ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια σε εσά για το έργο σας. Είμαι νέος βουλευτής βέβαια και νέος στην ε, Επιτροπή αυτή, αλλά έχουμε παρακολουθήσει όλοι ήδη από τα κράτη-μέλη μας την επιτυχία που είχατε στην ε, ε, διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας και την επιτυχία σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ενεργειακών προβλημάτων. Ένα σύντομο ερώτημα. Εγώ θεωρώ ότι ο κανονισμός για την ενέργεια <clears throat> περιλαμβάνει δύο πτυχές. Καταρχήν την εξασφάλιση της τροφοδοσίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις χώρες της Βαλτικής είναι πολύ σημαντικό διότι η προέλευση της ενέργειας για μας είναι κυρίως η Ρωσία και έχουμε προβλήματα με την ασφάλεια εφοδιασμού. Επομένως αυτό είναι το επόμενο ερώτημά μου, τι θα συμβουλεύσετε στον διάδοχό σας για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό της ενεργειακής ασφάλειας, ιδίως όταν πρόκειται από τη Ρωσία η ενέργεια. Κύριος Τούρμες. Κύριε Επίτροπε. Δεν ε, θα κάνω πολύ, δεν σας κάνω πολύ σε τέλος πάντων, αλλά όταν βγήκατε, όταν βγήκατε ε, επίτροπος, όταν οριστήκατε ο επίτροπος και ήρθατε εδώ, λέγανε όλοι πίμπαλς, ποιος είναι αυτός. Και όμως σήμερα είστε ένα από τους πιο ε, σεβαστούς Ευρωπαίους επιτρόπους και ο κύριος Ποτότσινγκ, ο οποίος ήταν ε, κάποιος άγνωστος ε, και εσείς είσαστε με μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη, διότι αποδείξατε ότι από το νέες, ε, με τις νέες χώρες μπορούμε να έχουμε κάποιους άγνωστους αλλά πάρα πολύ αποτελεσματικούς επιτρόπους. Δύο ερωτήσεις. Το εν, μια ερώτηση αφορά το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψη. Θα θυμόσαστε ότι όταν διαπραγματευόμεθα το, το σχέδιο ανάκαμψης κάναμε μια γραπτή δήλωση και θα ήθελα να ξέρω γιατί εμείς δεν πήραμε το πρόγραμμα ε, δράσεις για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα το Νοέμβριο έτσι όπως το είχαμε προβλέψει. Επίσης για την χρήση των ε, χρημάτων που δεν έχουν ε, δαπανηθεί. Το, η Κομισιό όταν υποβάλλει την έκθεση το 2010 για την εφαρμογή του κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 88 ε, θα μας παρουσιάσει και ε, τα χρήματα τα οποία δεν έχουν δαπανηθεί ε, και θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα να τα δώσουμε σε κάποια project για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Θα δώσετε κάποιε παρόμοιε συμβουλέ στο διάδοχό σας. Τελευταία ερώτηση. Μου είπαν ότι η Κομισιό θα υποβάλει νέα σενάρια για την ενέργεια μέσα στα πλαίσια το, του, της, της επόμενης ενεργειακής αναθεώρησης. Αυτά τα σενάρια θα τα ε, εξετάσει ο κ. Και ε, υπάρχει ένα ένα πρόσφατο σενάριο δικό του, το οποίο δεν σέβεται για καθόλου τους στόχους που είχαμε υιοθετήσει για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και στο παρελθόν. Και μου είπαν ότι ο κύριος Κάμπρος τώρα προτείνεται προτείνει ένα νέο επίσημο ευρωπαϊκό σενάριο όπου η Κομισιόν λέει ότι δεν θα σεβαστούμε τους στόχους του 2020 ούτε τους ε, στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ούτε τους ε, στόχους ε, για την, για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Ε, ήθελα να ξέρω εάν ε, αυτό υλοποιηθεί τελικά. Πιστεύω ότι είναι μια κατάχρηση, είναι μια σύγκρουση συμφερόντων, ε, είναι μια παραπλανητική, πολιτική που δεν πρέπει να εφαρμοστεί από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πάρα πολύ για, την, για τις πλήρεις εξηγήσεις που μας δώσατε για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ανάκαμψη και νομίζω ότι είναι και πολύ καλή στιγμή για να σας ευχαριστήσω για το ανοιχτό πνεύμα το οποίο δείξατε τα τελευταία πέντε χρόνια όταν μιλούσατε με τα μέλη αυτής της Επιτροπής και πραγματικά είχαμε πάρα πολύ ε, καλές σχέσεις ε, μεταξύ μας. Θα, σας, θα μας λείψετε πάρα πολύ. Σαν μέλος όμως της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης χαίρομαι ιδιαίτερα που αναλάβατε αυτό το χαρτοφυλάκιο γιατί χρειάζεται και πάρα πολύ δουλειά να γίνει για να προωθήσουμε και τις αναπτύξει ανανεώσιμε πηγές ενέργειας σε αναπτυσσόμενες χώρες. Πιστεύω ότι εξηγήσατε πάρα πολύ καλά για το πώς είναι δύσκολο να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό ε, μία ανοιχτή για το σχέδιο ανάκαμψη. και αυτό είναι αλήθεια. Όμως ε, ε, υπάρχει και μια ανησυχία για το πώς ε, δαπανώνται τα χρήματα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Βέβαια είναι καλό ε, γιατί τα, όλα τα χρήματα αυτά τα δαπανούμε για την ανάκαμψη και για όλα αυτά τα παράκτια, αιωλικά πάρκα κτλ. Αυτό το οποίο θέλω να ξέρω είναι ναι, ότι, δεν θα υπάρχουν άλλες καθυστερήσεις. Αναφερθήκατε επίσης και στη συνεργασία των κρατών μελών σε θέματα ανταγωνιστικότητας και θα πρέπει τα χρήματα αυτά όμως σίγουρα να δαπανηθούν γρήγορα. Τώρα, εάν υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις που ήδη υπάρχουν, κυρίως όσον αφορά τα σημεία διασύνδεσης, πώς ε, θα είμαστε σίγουροι ότι τα χρήματα αυτά δεν θα χαθούν, δεν θα παγώσουν τα κονδύλια και πώς θα χρησιμοποιηθούν με έναν αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο, κυρίως όσον αφορά την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα, ε, είναι, ε, θα έχει άμεσα αποτελέσματα στην, στην ανάκαμψη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω εν συντομία. Ήταν πάρα πολλά ερωτήματα. Θα έπρεπε κανονικά να, να δώσω μια πιο εκτενή απάντηση στην κυρία Γκιούρτς. Είναι γεγονός ότι οι χώρες της κεντροανατολικής Ευρώπης δεν έχουν σημεία, δεν έχουν κόμβους διασύνδεσης. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά το σχέδιο ανάκαμψης είναι το πρώτο εργαλείο αυτού του είδους. Μάθαμε πολλά από το πώς να το χρησιμοποιούμε και οι χώρες αυτές μάθανε πολλά επίσης και νομίζω το μελλοντικό μέσο για την ασφάλεια εφοδιασμού θα είναι ο κατάλληλος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα γιατί θα αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα ελλείψεων και το EPR, το πρόγραμμα αυτό ανάκαμψης, θα μπορέσει να είναι πιο επωφελές σε μια είναι περισσότερο μάλλον ένα εργαλείο που αντιμετωπίζει συγκεκριμένα την ενεργειακή κρίση, αλλά δεν είναι το πιο κατάλληλο εργαλείο για τα θέματα των κόμβων διασύνδεσης. Επίσης έχουμε προωθήσει το σχέδιο Smart Cities για την ενεργειακή αποδοτικότητα στους αστικούς χώρους και είναι απαραίτητο να έχουμε χρηματοδότηση για τα προγράμματα αυτά ενεργειακής αποδοτικότητας. Είναι κάτι το οποίο με την ευρωπαϊκή προώθηση θα επιτύχει πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούν να επιτύχουν μεμονωμένα τα κράτη-μέλη. Τι πρέπει να κάνει ο διάδοχός μου, όπως είπε η κυρία Χίμπνερ, Προφανώς δεν είναι μονάχα θέμα να έχουμε ένα ευχολόγιο. Θα πρέπει ο διαδοχός μου να είναι σε πολύ καλή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να είναι πάντα διαθέσιμος να ακούσει τις απόψεις των μελών της Επιτροπής Ενέργειας και Έρευνας. Είναι γεγονός ότι μπορεί να αποκλίνουν οι απόψεις, αλλά πάντα υπήρξε μια, ένας κοινός άξονας. Ζητήσαμε να υπάρχει μια μεγαλύτερη φιλοδοξία από την πλευρά της Κομισιόν πάντα στα θέματα της προσέγγισης για τα ενεργειακά θέματα. Και δύο θέματα μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Όπως είπε ο κ. Σόντι, μία πτυχή είναι οι καταναλωτές. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και στην πτυχή των καταναλωτών να δώσουμε μια μεγαλύτερη δυνατότητα εκ των κάτω προς τα άνω να διαρθώσουμε τον τομέα της ενέργειας και από την άλλη πλευρά φυσικά είναι και το θέμα της ευρωπαϊκής αντιμετώπισης. Να υπάρχουν οι διασυνδέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Αυτά τα θέματα θα πρέπει να αντιμετωπίσει, πιστεύω, ο διαδοχός μου, αλλά είναι πάρα πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για τον κύριο Σφόμποντα. Νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Σίγουρα εμείς θα προβούμε σε μια ανάλυση και θα επανέλθουμε με τις κατάλληλες προτάσεις. Είναι πολύ εύστοχο αυτό, η εύστοχη η ερώτησή σας για την κυρία Ποδηματά. Πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική υποστήριξη για όλα αυτά τα σχέδια που βρίσκονται στα ευρωπαϊκά μέσα. Τα σχέδια ευρωπαϊκού συμφέροντος λοιπόν θα εξακολουθήσουμε να τα υποστηρίζουμε στα συγκεκριμένα αυτά σχέδια που αναφέρατε και εσείς. Και φυσικά έχω δώσει εν μέρη μια απάντηση στο ερώτημα για το νέο μέσο το οποίο θα αφορά την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το θέμα της οριμότητος εδώ είναι κάτι το οποίο είναι μια προϋπόθεση. Έχουμε αναφέρει ότι τα χρήματα αυτά, μάλλον το σημείο, η χρονική στιγμή που θα είναι όριμα τα προγράμματα, εμείς δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε τα χρήματα πριν να οριμάσει ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο και γι' αυτό εμείς δεσμευτήκαμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα μέχρι το τέλος του 2010 για τα συγκεκριμένα προγράμματα που αναφέρατε. Κυρία Καρβάλιο, όλα αυτά τα οποία έχουν λειτουργήσει πολύ θετικά, έξι μείον ένα προγράμματα, μόνο ένα δεν ήταν από τα έξι δηλαδή έτοιμο, για τα έξι από αυτά τα προγράμματα εκτό από το ένα μπορούμε να δώσουμε τα χρήματα και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου και μας δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα <clears throat> να διαπραγματευτούμε καλύτερα για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής στην Κοπενχάγη. Για τον κύριο Χατζημαρκάκη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα κονδύλια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Εμείς προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε τις ενέργειές μας σε συγκεκριμένα σχέδια και σε διασυνδέσεις, γιατί αυτό θα βελτιώνει την κατάσταση. Αλλά δεν πρόκειται μονάχα για μεγαλύτερη ανάπτυξη στα υπεράκτια αεολικά πάρκα. Εγώ ε, σας παροτρύνω να πάτε να δείτε ένα πρόγραμμα το οποίο έγινε στην Εστίν σε απόσταση 65 χιλιόμετρων από τις Βρυξέλλες, ένα αιωλικό πάρκο 7 ΜΒ. Υπήρξε πραγματικά ενδιαφέρον σε τοπικό επίπεδο από τη νέα τεχνολογία και όχι απλώς μια συντηρητική αντιμετώπιση και πιστεύουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιδιαίτερα όλα αυτά τα σχέδια. Κανείς δεν θα πίστευε ποτέ ότι θα έχουμε τουρμπίνες 7 ΜΒ σε, σε μια τοποθεσία όπως αυτή στο Βέλγιο. Υπάρχει μεγάλη δυναμική λοιπόν σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση των αιωλικών πάρκων. Αν θα έχει ο επόμενος επίτροπος αρκετές εξουσίες δεν θα έχει ακριβώς όλες αυτές τις, ε, τις ε, εξουσίες που είχα εγώ και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει και σύγκρουση συμφερόντων από την άποψη αυτή. Είναι καλό ότι ο Επίτροπος για τις για την ενέργεια δεν θα έχει αυτές τις πτυχές, τις πτυχές του ανταγωνισμού και των κρατικών επιδοτήσεων για τον άνθρακα. Νομίζω ότι είναι καλύτερη η θέση του επερχόμενου λοιπόν επιτρόπου. Το ερώτημα του κυρίου Όντι. Υπάρχουν κάποια φιλοσοφικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε προφανώς, αλλά σε σχέση με τα θέματα ενέργειας και το Κοινοβούλιο. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία μας δίνει η συνθήκη. Αλλά έχουμε κάποιες δυνατότητες πρωτοβουλίες για την ενεργειακή αποδοτικότητα, για την προστασία των καταναλωτών και όλα αυτά νομίζω ότι αυτά είναι θετικά μηνύματα τα οποία μπορούμε να δώσουμε στους Ευρωπαίους για τα θέματα της ενέργειας. Στο παρελθόν ήταν απλώς σαν να κηρύττουμε ε, από άμβονος. Αυτή τη στιγμή με το γεγονός ότι έχουμε δώσει αυτή τη χρηματοδότηση στα 4 δισεκατομμύρια δείχνουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους για να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες που είναι προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το ερώτημα για την ε, Βαλτική. Έχουμε ένα σχέδιο για ανάπτυξη διασυνδέσεων στη Βαλτική. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το πρόγραμμα και να το εφαρμόσουμε και για τον ηλεκτρισμό και για το φυσικό αέριο και να συνεχίσουμε την εκτέλεση αυτού του προγράμματος όπως όπως προβλεπόταν. Για τον κύριο Τούρμες, το σχέδιο δράση για την ενεργειακή απόδοση ήταν έτοιμο να συζητηθεί από την ε, Κομισιόν, αλλά λόγω της καθυστέρησης με την κύρωση της ε, Συνθήκης Λισαβόνας θα το αναλάβει το επόμενο σώμα των Επιτρόπων. Δυστυχώς υπάρχουν παρεμβολές από κάποιο κινητό τηλέφωνο. Γι' αυτό δεν ενεκρίθη από το Σώμα των Επιτρόπων, αλλά είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατό από, το νέο, από τη νέα Κομισιόν. Για το ρυθμιστικό πλαίσιο. Έχουμε ένα πρωτόκολλο το οποίο εγώ δεν έχω λησμονήσει. Θα σας υπενθυμίσω μια φράση για το θέμα αυτό, ότι μετά από την περάτωση των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για τις διασυνδέσεις, που αναμένεται να γίνουν στο τέλος του 2010 θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα για την απορρόφηση του προπολογισμού. Την άνοιξη του 2010 η Κομισιόν θα δώσει την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 28 του κανονισμού και μέχρι τότε η Κομισιόν θα έχει αξιολογήσει διάφορες εναλλακτικέ λύσεις σε σχέση με την δαπάνη πιστώσεων υποχρεώσεων που δεν θα έχουν εκταμιευτεί με ένα τέτοιο τρόπο που να επιτρέψει την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού για το EPR. Και αυτό περιλαμβάνει το πρωτόκολλο για το οποίο συμφωνήσαμε. Δεν έχουμε ξεχάσει λοιπόν τη συμφωνία που έχουμε κάνει μαζί σας. Για τα εναλλακτικά σενάρια. Είναι ένας δύσκολος ανηφορικός αγώνας. Πολλές φορές είναι δύσκολο να καταλάβω τη λογική αυτών που εκπονούν τα σενάρια. Είναι εμπειρογνώμονες αυτοί, αλλά για μένα ο στόχος του 20% εξακολουθεί να είναι ο προεξάρχων. Πρέπει και αυτοί λοιπόν που εκπονούν τα διάφορα σενάρια να τροποποιήσουν τη μεθοδολογία τους. Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν την εργασία, αλλά η Κομισιόν δεν μπορεί να δεχτεί κανένα σενάριο το οποίο δεν επιτυγχάνει το στόχο του 20% μείωσης ε, των εκπομπών το 2020. Αν μειώνει ακόμα περισσότερε εκπομπέ, βεβαίω μπορούμε να το εξετήσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε τίποτα που έχει μείωση κάτω από το 20%. Γι' αυτό εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα σενάρια θα υπακούν σε αυτές τις προδιαγραφές για το μέλλον. Για την κυρία Χολ, νομίζω ότι καταδείξαμε ότι αντιμετωπίζουμε σωστά αυτό το θέμα. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι είναι <clears throat> απαραίτητο η Επιτροπή Βιομηχανίας να είναι σε επαφή με το προσωπικό, με την ε, γενική μου διεύθυνση όσο δυνατόν συχνότερα, γιατί μαθαίνουμε κάνοντας. Όταν πρόκειται λοιπόν για την υπογραφή των συμβάσεων, μπορούν να προκύψουν προβλήματα. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Εγώ θεωρώ ότι είναι θετική κατάσταση και δεν υπάρχουν ελοχεύοντες κίνδυνοι όπως είναι τώρα τα πράγματα ότι δεν θα εκταμιευθούν τα χρήματα αυτά ή ότι θα χαθούν. Είναι πολλά όμως τα προγράμματα τα οποία θα εγκριθούν κάτω από ορισμένε προποθέσει. Αυτό είναι ο δυναμικό χαρακτήρα τη διαδικασία και εμεί θέλουμε να τονίσουμε ότι θα έχουμε αυστηρά κριτήρια και ποιοτικά κριτήρια. Θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον. Θέλω να σα ευχαριστήσω λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τι πληροφορίε σας, για την προθυμία που επιδείξατε τα τελευταία πέντε χρόνια να έρθετε να κουβεντιάστε μαζί μας στην Επιτροπή μας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και είμαι σίγουρη, σίγουρος ότι και οι συνεργάτες έχουν την ίδια άποψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Äh, λοιπόν, προχωρούμε στο επόμενο θέμα για την ασφάλεια του αφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Η έκθεση του κυρίου Βιντάλ Κουάδρας υπάρχει, ε, την έχετε στη διάθεσή σας. Θα του δώσουμε το λόγο για να μας κάνει ως συγητής μια κάποια εισαγωγή. Ε, ενδεχομένως να υπάρχουν βεβαίως ερωτήσεις τις οποίες θα πρέπει να απαντήσει αλλά βρισκόμαστε στο στάδιο εξέτασης του σχεδίου έκθεσης Βιντάλ Κουάδρας. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε τώρα να έχουμε και μία ανταλλαγή απόψεων επί τη βάση ενός κειμένου που είναι η πρότασή μου, το σχέδιο εκθεσής μου και όπως θα παρατηρήσουν και οι συνάδελφοι, περιλαμβάνει στοιχεία από πολλές συζητήσεις και προσωπικές συζητήσεις που κάναμε με πολλά μέλη της Επιτροπής μας. Επίσης, τα απορίσματα των επαφών με τους εμπλεκόμενους τομείς, συζητήσεις με τους κοιόδης εισηγητές επαφές με την Κομισιόν. Ως εκ τούτου, η ελπίδα μου είναι ότι οι τροπολογίες που θα προτείνω εγώ σε αυτό το στάδιο, ότι πράγματι αντικατοπτρίζουν την καταπλειοψηφία θέση της Επιτροπής μας. Τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος μου, αυτό το οποίο ελπίζω ότι θα μπορέσω να επιτύχω μετά από την ε, σφιγμομέτρηση κάπως που έκανα ε, σε σχέση με τα θέματα αυτά μεταξύ των συναδέλφων και τις επαφές μεταξύ ημού και αυτών. Θέλω να αναφέρω μερικές από τις πιο σημαντικές τροπολογίες τώρα και, στα σημεία, και τα σημεία που αναφέρονται. Καταρχήν υπάρχει ο ρόλος των επιχειρήσεων. Είχαμε πει και στο παρελθόν <clears throat> ότι το κείμενο δεν συντεριάζεται απόλυτα ούτε με τις δηλώσεις της Κομισιόν ούτε με αυτά που λέμε στι αιτιολογικέ σκέψει. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση σε πολλά επίπεδα, και ένα από αυτά τα επίπεδα είναι η αγορά, αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο κείμενο, να αντανακλάται με έναν τρόπο που θα είναι σαφέ και γι' αυτό εγώ έχω εισαγάγει ορισμένε τροπολογίε σε διάφορα σημεία, των οποίων ο στόχο είναι να υπογραμμίσω ότι τα μέτρα τα οποία δεν είναι μέτρα στήριξη τη αγορά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο σε ακραίες συνθήκες σαν τελική δυνατότητα αντιμετώπισης. Θα πρέπει να αφήσουμε τον κύριο ρόλο στην αγορά. Δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να αναφέρω και το οποίο ίσως δημιούργησε ανησυχίες σε πολλούς συναδέλφους είναι το θέμα της κατανομής του κόστους κατασκευής υποδομών σε κράτη-μέλη όταν από αυτές τις υποδομές ωφελείται άμεσα ένα άλλο κράτος μέλος. Εδώ έχω προτείνει μια τροπολογία η οποία έχει να κάνει με αυτή την κατανομή του κόστους και έχω συνδέσει αυτή την τροπολογία με αυτά τα οποία είχαν ήδη συμφωνηθεί στο τρίτο πακέτο της εσωτερικής αγοράς και της ενέργειας, ότι πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων και να εφαρμοστεί ένα κριτήριο αναλογικότητας σε ό,τι αφορά την κατανομή του κόστους. Ένα τρίτο θέμα αφορά τις αμφίδρομες ροές. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικότητα σε ό,τι αφορά την αμφίδρομη ε, ροή όταν πρόκειται για προσφορά πρόσθετης ασφάλειας σε ό,τι αφορά την ενεργειακή τροφοδοσία. Όχι κάτι που θα είναι υποχρεωτικό. Και τέταρτον, μου φαίνεται λογικό να προτείνω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να προβεί σε μια ανάλυση κινδύνων και να έχει ένα σχέδιο προβλέψεων για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο πρόληψης το οποίο θα εξασφαλίσει ότι τα εθνικά σχέδια θα είναι συγκλίνοντα θα είναι συνεκτικά μεταξύ τους και το σχέδιο αυτό θα πρέπει επιπλέον να κάνει συστάσεις προς τα κάτι μελη προς την κατεύθυνση αυτή. Ένα πέμπτο σημείο, η ομάδα συντονισμού θα πρέπει να συμμετάσχει περισσότερο σε στιγμές κρίσης, θα πρέπει να δίνει συστάσεις προς όλους τους εμπλεκόμενους, είτε για να καθοριστούν οι περιοχές όπου είναι πιο απαραίτητη η περιφερειακή συνεργασία, είτε για την εκπόνηση σχεδίων πρόληψης. Μια έκτη πτυχή που θέλω και αυτή να αναφέρω είναι αυτή των κατοφλίων για να θεωρηθεί ότι σοβεί πράγματι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ρήτρε και πρόνοιες που αφορούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που είναι ιδιαίτερα εντοπισμένες στο χώρο. Θα πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρχει κοινοτική παρέμβαση σε συνθήκες οι οποίες είναι και πιο διαφοροποιημένες. Δηλαδή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι μπορούν να προκύψουν καταστάσεις που σε τοπικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα σοβαρές, αλλά σε ένα γενικό κοινοτικό πλαίσιο βάσει των ποσοτικών κριτήριων τα οποία χρησιμοποιούμε φαίνονται ίσονα προβλήματα. Αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε να μην αντιμετωπίζονται λόγω του συνολικού χαρακτήρα τους, ενώ είναι πολύ σημαντικές σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά από μια ευρωπαϊκή άποψη, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και την απαραίτητη αλληλεγγύη. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω και μια σειρά από τροπολογίες που τροποποιούν διάφορες πτυχές του κανονισμού, <clears throat> όπως παραδείγματος χάρη η συμπερίληψη του αντικτύπου στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάγκη να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε τις διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών και την ανάγκη να υπάρξει σε μέσο και μακροπρόθεσμο επίπεδο ένα σχέδιο δράσης για την διαφοροποίηση των πηγών ε, εφοδιασμού και των διαδρομών εφοδιασμού με ιδιαίτερο, ε, ιδιαίτερη έμφαση στους σταθμούς αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου. Υπάρχουν ορισμένα θέματα, αγαπητοί συνάδελφοι, τα οποία ακόμα δεν τα έχω αντιμετωπίσει και υπογραμμίζω το μέχρι στιγμής. Ένα από αυτά τα θέματα είναι ο ορισμός του τι είναι οι προστατευόμενοι πελάτε και το άλλο είναι ο κανόνας νήμιον ένα σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Όπως είπα προηγουμένως, είναι θέματα τα οποία είναι μεν σημαντικά μέσα στον κανονισμό αυτό που οδηγούν σε άμεσες επιπτώσεις για τις επενδύσεις οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και επίσης για τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλίσουμε την τροφοδοσία σε ενέργειες. Αλλά εγώ δεν έχω αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά ακόμα γιατί πιστεύω θα πρέπει να συζητηθούν σε μεγαλύτερο βάθος. Με τους και με το σύνολο των συναδέλφων στην Επιτροπή μας και ξέρω επίσης ότι και η Κομισιόν επεξεργάζεται τα θέματα αυτά. Ως εκ τούτου δεν έχουν οριμάσει οι προβληματικές για τα θέματα αυτά, ώστε να μπορέσω να μεταφέρω στην Επιτροπή μας μια συγκεκριμένη πρόταση. Θα ήθελα η πρόταση αυτή να προέλθει μετά από μια συμφωνία με όλους τους εμπλεκομένους. Για τους προστατευόμενους πελάτες. Αυτό το οποίο θα ήθελα να έχουμε είναι να υπάρξει μια συμφωνία όλων μας σε σχέση με ένα φάσμα κριτηρίων τα οποία θα σέβονται τα κράτη-μέλη εάν θέλουν να περιλάβουν και κάποιους άλλους καταναλωτές πέραν των οικοκυριών. Γιατί ορισμένοι έχουν μια διασταλτική ερμηνεία και άλλοι μια πολύ στενή ερμηνεία. Ζητούν ορισμένοι να περιληφθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι 80% της ευρωπαϊκής οικονομίας. Άλλοι λένε γιατί όχι τα σχολεία, γιατί όχι τα νοσοκομεία, γιατί όχι οι πυροσβέστες, γιατί όχι η αστυνομία. Νομίζω λοιπόν ότι ένας εξαντλητικός κατάλογος δεν είναι η καλύτερη λύση, γιατί το κάθε κράτος έχει ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Αν προσπαθήσουμε να έχουμε ένα εξαντλητικό κατάλογο, πάντα θα εξέφευγαν ορισμένε καταστάσει που είναι σημαντικέ για ορισμένα κρατημέλη. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια σειρά γενικών κριτηρίων, τα οποία να είναι εύκαμπτα, να μπορούν να προσαρμοστούν στι συνθήκε τι ιδιαίτερε των κρατών μελών, να έχουν χαρακτήρα αποτελεσματικό αλλά και εύκαμπτο. Σε σχέση τώρα με τον κανόνα νη 1 παραμένουν ακόμα αστάθμητα στοιχεία σε σχέση με την εφαρμογή του και το σχήμα το οποίο θα πρέπει να διέπει αυτόν τον κανόνα. Εγώ νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα, ένα καλό κριτήριο να διατηρήσουμε τον κανόνα αυτό τον νη 1 και να τον βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Στη χώρα μου λειτουργεί πολύ καλά ο κανόνας αυτός. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εξευγενήσουμε λίγο περισσότερο αυτόν τον κανόνα για να είναι ένα εργαλείο εργασία το οποίο να είναι ομοιόμορφα αποτελεσματικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντα όμω και πάλι υπόψη τι διαφορέ οι οποίε υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών μα. Είναι ένα ιδιαίτερα τεχνικό θέμα και θα να προσκαλέσω όλου του συναδέλφου οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμβάλλουν για τη διαλεύκανση αυτού του προβλήματο. Η δική μου πρόταση θα ήταν να ενισχύσουμε τι ε, ρήτρες αυτές οι οποίες καθορίζουν βάσει ποιων κριτηρίων μπορούμε να εφαρμόσουμε τον κανόνα του νη και να θεωρήσουμε ότι έχει επιτευχθεί η εφαρμογή αυτού του κανόνα και συγχρόνως να προσθέσουμε στο πρώτο παράτημα με νέες πρόνοιες που και με την εξάλληψη ορισμένων προδιαγραφών για την τροφοδοσία που δημιουργούν σύγχυση γιατί είναι διαφορετικό το θέμα των υποδομών, να μπορούν να λειτουργήσουν ανελιπώς οι υποδομές, αυτή είναι η προσέγγιση από την πλευρά των υποδομών, και άλλο θέμα είναι οι προδιαγραφές εφοδιασμού. Σε μια κατάσταση κρίσης όλοι οι προστατευόμενοι πελάτες θα πρέπει να καλυφθούν. Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες, τις οποίες δεν θα πρέπει να συγχαίουμε μεταξύ τους, γιατί αυτό θα μας οδηγούσε σε μια πλήρη σύγχυση. Ο κανόνας λοιπόν είναι μειον <clears throat> για τις υποδομές. Είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε μακροπρόθεσμο επίπεδο γιατί απαιτεί τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, απαιτεί ένα σχεδιασμό πιο μακρόπνο. Αυτή είναι μία λοιπόν προσέγγιση. Ενώ η άλλη προσέγγιση είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ότι τη στιγμή που ξεσπάει μια κρίση θα πρέπει να έχουμε καλύψει μια σειρά από προστατευμένων πελατών και χρηστών τη ενέργεια. Αυτά ήθελα να πω λοιπόν κύριε Πρόεδρε σε σχέση με την πρώτη αυτή πρόταση την οποία παρουσιάζω, το πρώτο σχέδιο εργασία. Θα πρέπει να ακολουθήσει λοιπόν μια συζήτηση και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και ιδίως τους σκιώδεις εισηγητές για τη βοήθεια που μου έχουν δώσει μέχρι στιγμής για την εκπόνηση αυτού του σχεδίου έκθεση και προφανώ εγώ θα συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί του για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε, ήταν ε, πάρα πολύ ε, καλή παρουσίαση. Δέκα ομιλητές έχω στο κατάλογο, αλλά έχουμε και άλλα θέματα στην ημερήσια διάδειξη. Επαναλαμβάνομαι λοιπόν και σε ζητώ συγκεντρωθείτε και πάλι στα βασικά, διότι ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε στην έκθεση αυτή του κυρίου Βιντάλ Κουάδρας και ζήτησε και ο εισηγητής να υποβάλλετε γραπτά σχόλια αν έχετε. Ο κύριος Φόμποντα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Βινταλ για την ε, δουλειά που έκανε και την παρουσίαση. Είναι πάρα πολύ καλό να ε, τονιστεί το θέμα των εταιριών αερίου και το θέμα του συντονισμού. Αυτά τα χαιρετίζουμε. Επίσης η πρόταση ε, τον, την περιγραφή την επακριβή της κοινοτικής έκτακτης ανάγκης αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ καλή διότι μέχρι τώρα δε, σαφής ορισμός δεν είχε δοθεί για το emergency που λέγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το άλλο θέμα για τη διαφοροποίηση τώρα Ίσως εκεί χρειαστεί να ζητήσουμε και άλλες πληροφορίες από την Κομισιόν αν μιλώντας για διαφοροποίηση μιλούμε μονάχα για πηγές προμήθειας, πηγές εφοδιασμού είναι διαφορετικά τα πράγματα ε, θα ήθελα εδώ μερικά σχόλια. Τέταρτο θέμα για την εφαρμογή των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Ίσως θα έπρεπε να πούμε ότι μετά από τρία χρόνια θα πρέπει να γίνει μια ενδιάμεση έκθεση για να διαπιστωθούν τα προβλήματα. Στα πέντε χρόνια θα πρέπει να έχουν διορθωθεί. Τώρα, για την την, τα δεδομένα και την ε, διαβίβαση δεδομένων ε, και συγκέντρωση των στοιχείων αυτών εάν τα δεδομένα αυτά είναι σωστά συγκεντρωμένα και μπορεί να τα επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Κομισιόν εντάξει εδώ όμως πρέπει να προσέξουμε από εκεί και πέρα ε, για την άλλη πρόταση που κάνει ο κύριος Βιντάλ Κουάντρας θα πρέπει να ε, ε, να ξαναδούμε λιγάκι το θέμα των διαφορών μεταξύ γενοτονικών κρατών μελών ε, και πώς θα μπορεί να επέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκεί τώρα από εκεί και πέρα ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι στις διαφορετικές χώρες ε, υπάρχει διαφορετική ευελιξία και ίσως εδώ πρέπει να επέμβουμε, θα το δούμε ε, αυτό στις επόμενες συζητήσεις μας. Τώρα από εκεί και πέρα ε, πρακτικά, δεν ξέρω όλα Ξέρω από το Συμβουλίο, ίσως να μπορέσουμε ε, να ε, τελειώσουμε μετά την πρώτη ανάγνωση. Πάντως νομίζω ότι η έκθεση του κυρίου Βιντάλ Κουάδρα σε πολύ καλή βάση για μελλοντική συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ Σιμάνσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η, ο, η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και οι παρουσίες που έκανε ο συγητής ε, πολύ καλή νομίζω είναι σημαντικό το ότι ζητεί ο εισηγητής καλύτερο συνταγισμό, καλύτερη συνεργασία ε, αυτά τα χαιρετίζουμε για το θέμα της διαφοροποίησης ίσως θα πρέπει να υπάρχει και ένας ε, μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης κάπου πρέπει να το προσθέσουμε και αυτό βεβαίως οι αγορές είναι αυτές οι οποίες θα αντιδράσουν πρώτες και θα ε, προσπαθήσουν να βοηθήσουν οπότε ίσως να μην χρειάζεται να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου απέτυχε αν θέλετε η αγορά να αντιδράσει ή να διορθώσει ορισμένα πράγματα. Τώρα υπάρχουν βεβαίως και τα εθνικά σχέδια και σχετικά θα πρέπει να πούμε ότι θα υποστηριχθούν μοναχά εκείνες οι δράσεις οι οποίες έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Δεν προσπαθώ τώρα να περιορίσω το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσεως. Ε, εάν ε, γίνουν κάποια πράγματα τα οποία αποβαίνουν ή ενδέχεται να αποβούν προς ζημία ε, κάποιας ε, χώρας ε, βεβαίως πρέπει να ε, παρέμβει η Επιτροπή επίσης για το, το κανόνα του εν μείον ένα είμαστε υπέρ της επέκταξης του κανόνα αυτού και όσον αφορά τώρα την αντίστροφη ροή πράγματι είναι γεγονός ότι δεν χρειάζεται πάντοτε αλλά χρειαζόμαστε τις αντίστροφες ροές σε γενικές γραμμές ο, ο ενδιαφερόμενος όμως η ενδιαφερόμενη ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να μπορεί να ζητήσει διακοπή αυτής της αντίστροφης ροής. Εγώ νομίζω όμως ότι θα πρέπει, ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα αυτό τώρα από εκεί και πέρα για την ε, έκτακτη ανάγκη οποιαδήποτε μέτρα πάρουμε σχετικά δεν θα πρέπει να αποβούν εις βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος των δράσεων που προβλέπουμε για τις κλιματικές αλλαγές. Όσον αφορά τα δεδομένα και τα σχετικά προβλήματα νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες δεδομένων τις οποίες θα πρέπει να διατηρήσουμε ίσως όχι άλλες διότι αν κάποια δεδομένα αποκριστούν τότε η Κομισιόν μπορεί να μην έχει τα στοιχεία που της χρειάζονται να μπορέσει να αντιδράσει Ευχαριστώ πολύ Κύριε Στούρμα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Βιδάλ Κουάδρας. Είναι πολύ καλή η εργασία αυτή την οποία μας έχετε παρουσιάσει και δεν με εκπλήσει, διότι είσαστε ένα από τους πραγματικούς, από τους πραγματικούς εμπειρογνώμονες στο θέμα αυτό. Εξού και θα επικεντρώσω την προσοχή μου σε κάποια θέματα, σε κάποια σημεία, για τα οποία θα μπορούσα να ζητήσω να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Καταρχάς πρέπει να είναι σαφές ότι τα εργαλεία της αγοράς και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι το καλύτερο φάρμακο και θα πρέπει να το ενδυναμώσουμε, να ενδυναμώσουμε την τυχή αυτή στο κείμενο. Μετά χρειαζόμαστε έναν ισχυρό ρόλο για τους ρυθμιστέ. Ε, ε, ρυθμιστές. Αυτοί οι ρυθμιστές θα μπορούσαν ε, να χρησιμοποιηθούν και από τα κράτη-μέλη τα οποία δεν θέλουν ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά του φυσικού αερίου για να μειωθεί η ισχύ των ρυθμιστών αυτών στον τομέα του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ενδυναμωθούν όμω. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία έτσι ώστε να εκπονήσουν τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης. Διότι τα άτομα αυτά γνωρίζουν καλύτερα ποια είναι τα σημεία ε, ισορροπίας ανάμεσα στην λειτουργία της ιδιωτικής αγοράς και την ενεργειακή ασφάλεια. Εξού και οι εθνικοί ρυθμιστές θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο. Όταν μιλάμε για έκτακτη ανάγκη, θα και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι και η κρίση η περσινή μας το έδειξε ότι ας πούμε παραδείγματος χάρη η Ιταλία αποφάσισε να κλείσει όλη τη την αγορά. Η Σλοβενία και η Σλοβακία προσπάθησαν να πάρουν φυσικό αέριο από την Γαλλία μέσω της Ιταλίας και αυτό τους πήρε τρεις εβδομάδες διότι η Ιταλία αποφάσισε να κλείσει τελείως τους αγωγούς για την διέλευση. Επομένως αυτού του είδους εθνική σκέψη, αποκλειστικά εθνική σκέψη δεν βοηθάει. Όταν υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη θα πρέπει να είναι σαφής ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένα σαφής ρόλος ε, που θα αφορά την περιφερειακή συνεργασία. Η περιφερειακή διάσταση, η περιφερειακή συνεργασία είναι μια πτυχή που πρέπει να ενδυναμωθεί στο κείμενο. Η Εσθονία, η Λιθουανία και η Λετωνία συνεισφέρουν ε, ε, και δημιουργούν ούτως ή άλλως μία αγορά αυτές οι τρεις χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ελλάδα. Εάν δείτε τους αγωγούς, εάν δείτε το, τις δομές για το υγραέριο, ε, θα ήταν παράλογο οι χώρες αυτές να μην έχουν περιφερειακά ε, προγράμματα για να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες και όχι καν εθνικά προγράμματα. Και στην, ε, στην υπάρχει και ένα εξάρτητο φόρουμ που και εκεί πιστεύω θα πρέπει να εκπονηθούν ε, τέτοιου είδου σχέδια έκτακτης ανάγκης. Τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε την διαφάνεια. Τη χρειαζόμαστε. Διότι αν η Κομισιό δεν έχει τις απαραίτητες πληροφορίες ε, από πλευρά των κρατών μελών και αν, και και το, και αν δεν υπα, δοθούν πληροφορίες στο Συμβούλιο, πώς μπορεί ένας τυφλός να μας οδηγήσει για να βγούμε από την κρίση. Εξού και πιστεύουμε ότι η κρίση, η, κρίση λέω, η Κομισιόν χρειάζεται πληροφορίες για να βγούμε από την κρίση. θα πρέπει γενικότερα να υπάρξουν ε, επενδύσεις και επενδύσεις γρήγορα. Γιατί ε, πιστεύουμε ότι ε, οι επενδύσεις αυτές θα αποδώσουν. Τώρα, για τα θέματα του 1-1, του νήμιον 1, συγγνώμη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ περίπλοκο επίσης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο Απευθύνω μια ερώτηση στην Κομισιό. Αν κατάλαβα καλά, η Κομισιό έχει προχωρήσει σε ανταλλαγές ε, πληροφοριών ε, με την Eurogas και όλες τις εταιρείες που προμηθεύουν ε, φυσικό αέριο. Είναι δυνατόν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου ή αρχές Ιανουαρίου πριν υποβάλουμε εμείς τις τροπολογίες θα μπορούσε η αρχες ιανουαριου πριν υποβαλουμε μεχρι τις τροπολογιες θα μπορουσε η κομισιο να μας υποβάλει ένα κείμενο ένα, που να λέει τι χρειάζεται να αλλαγεί να αλλάχθεί συγγνώμη, σε σχέση με την πρώτη σας πρόταση. Γιατί εμείς ε, σαν βουλευτές πρέπει να τα μελετήσουμε όλα αυτά, δεν τα καταλαβαίνουμε. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Βόμποντα, δεν πρέπει να ε, προκαλέσουμε στρέβλους του ανταγωνισμού. Διότι αν έχουμε μια εταιρεία η οποία επιτρέπεται να κάνει μια επένδυση σε ένα κράτος μέλος όπου προστατεύεται το φυσικό άριο και από την άλλη πλευρά ε, δεν θεωρηθεί αυτή η εταιρεία ευάλωτος πελάτης, ε, ε, ε, τι θα γίνει, δεν δημιουργείται μια στρέβλωση. Τώρα, όσον αφορά την αλληλεγγύη, πρέπει να, η αλληλεγγύη να εμφανίζεται και πρακτικά και όχι μόνο θεωρητικά. Και υπάρχει μια πρόσφατη συμφωνία ανάμεσα σε μια πολωνική εταιρεία και την και Gazprom, και την Gazprom και πραγματικά μου εκπλήσει το, με εκπλήσει το γεγονός ότι ενώ οι πολιτικοί μας ε, έβλεπαν με ιδιαίτερη καχυποψία την Gazprom και δεν είχαν καλά λόγια να πούν για αυτήν, ε, η, πλειοψηφία του φυσικού αερίου στην Πολωνία προέρχεται από εκεί. Και ε, γίνεται μια προσπάθεια να εισαχθεί μια ρήτρα στη συμφωνία που έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μήπως θα μπορούσε η Κομισιόν να μας το διευκρινίσει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ τους, ε, ε, για την παρέμβαση σας και σας παρακαλώ να είστε λακωνικοί γιατί δεν θα προλάβουν όλοι να μιλήσουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω την εξαιρετική δουλειά που έκανε ο Ισπανός συνάδελφος. Η σχέδια, το σχέδιο έκθεσης του ε, ανταποδίδεται πλήρως στις προσδοκίες των πολιτών μας μετά την κρίση την περσινή στο το, ε, τομέα του φυσικού αερίου που έθεσε σε κίνδυνο την ε, ασφάλεια εφοδιασμού της κοινότητας. Θα ήθελα να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. Καταρχάς, ε, πώς ορίζουμε τους, τους φορείς, ε, ε, τους αρμόδιους φορείς και λέγεται εδώ ότι οι αρμόδιοι αυτοί φορεί θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από το κράτο. Ήθελα να υπενθυμίσω όμω ότι η προμήθεια σε φυσικό αέριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ε, θέμα αρμοδιότητα των κρατών μελών και θα πρέπει να αναθέσουμε την, ε, την, την, τα θέματα αυτά της προμήθειας στις εθνικές αρχές. Επίσης μιλάμε για ανεξάρτητες ε, αρχές ε, που φορείς της αγοράς. Δεν το διευκρινίσουμε αυτό. Επίσης ο ευάλωτος καταναλωτής, ο, ευάλωτος, ο πελάτης. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό αφορά τα νοικοκυριά και αν το αποφασίσει, τα κράτη, το αποφασίσει το κράτη-μέλη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα νοσοκομεία, τα σχολεία κτλ. Συμφωνούμε να προστατευτούν τα νοικοκυριά, δεν έχουμε καμία αντίρρηση, αλλά για τις άλλες κατηγορίες που αναφέρονται εδώ, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κόστος που συνεπάγονται οι συμπληρωματικές επενδύσεις για να προμηθεύσουμε και να εφοδιαστούν οι εταιρείε αυτές. Το κόστος αυτό για τον καταναλωτή, το οποίο, ο θα πρέπει να πληρώσει μετά την αύξηση των τιμολογίων του φυσικού αερίου. Επομένως, ναι με να υπάρχει μια διεύρυνση των προστατευμένων πολιτών, όμως αφού γίνει μια, συμπληρω... μια ενδελεχής μελέτη του κόστους και ωφέλου και μετά από, συνδια... από διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι γεγονός ότι ο κανονισμός αυτός είναι ιδιαίτερα επίκαιρος και νομίζω ότι η δουλειά που έκανε ο εισηγητής μας και οι τροπολογίες του έχουν μεγάλη σημασία. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι χρειαζόμαστε μια ενιαία αγορά φυσικού αερίου στην οποία να έχουν πρόσβαση όλες οι εταιρείες. Είναι γεγονός ότι πρέπει να δούμε και τι γίνεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αλλά νομίζω ότι τα σχέδια έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να ορίζονται αναπεριφέρεια περιφερειακά και επίσης θα πρέπει να δούμε ότι είναι πολύ σημαντική η διασύνδεση και με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας η κατάσταση στις βαλτικές χώρες μάλλον στη Λιθουανία είναι εξαιρετική και ο κανόν είναι ιδιαίτερα ιδιαίτερη και ο κανονισμός αυτός ε, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με κάποιους περιορισμούς δεν, στην Λετωνία ε, παραδείγματος χάρη υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες αποθηκεύσης αυτά τα χρονοδιαγράμματα εδώ των έξι μηνών ε, είναι πολύ σύντομα κατά την άποψή μας και γι' αυτό που ελέγχθη προηγουμένως αν αποκοπούμε από την Gazprom τότε τελικά δεν θα έχουμε καθόλου φυσικό αέριο. Θα θυμάστε τα, το τι συνέβη το Γενάρη του 2009 ο αγωγός Ντρούστα έκλεισε και με αυτή την έννοια δεν είχαμε φυσικό αέριο και άλλα δεν είχαμε και, και καμία σύνδεση με την αγορά φυσικού αερίου. Γι' αυτό τονίζω ότι πρέπει να έχουμε μια ενιαία αγορά στο οποία να έχουν πρόσβαση όλα τα κράτη-μέλη. θα έπρεπε να υπάρχει ένας αγωγός από τη Βαλτική μέσω της Πολωνίας μέχρι την Αυστρία για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι το δεν ξέρουμε αν η Ρωσία θα τι θα κάνει η Ρωσία με τον Nord Stream και δεν ξέρουμε κατά πόσον θα μπορούσε, θα υπάρξει αν θέλετε παράκαμψη προς το Καλίνιγκραντ εν η περιπτώσει οι χώρες της Βαλτικής μπορεί να ε, ε, έχουν εναλλακτική δυνατότητα εφοδιασμού ε, εξαρτώμεθα συνάδελφοι από το ρωσικό αέριο ε, αυτό είναι γεγονός και επανέρχομαι και τονίζω ότι οποιαδήποτε ενιαία αγορά φυσικού αερίου πρέπει να προβλέπει ίση ε, πρόσβαση για όλους. Πρόεδρος, ναι, έχουμε πλήρη κατανόηση για το ότι ακρηγορήσετε δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι πραγματικά έχετε μεγάλο πρόβλημα. Uh, well, uh, Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το θαυμάσιο έργο του. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κύριε Βιδάλ Κουάδρας, ότι υποστηρίζω την προσέγγιση σας. Το πρώτο το οποίο θα ήθελα να πω και θα ήθελα να χαιρετήσω είναι το θέμα της διαφοροποίησης των διαδρόμων εφοδιασμού με φυσικό αέριο και των πηγών εφοδιασμού. Είναι ένα κεφαλαίωδες θέμα για μένα και χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος ε, Βιδάλ Κουάδρας το διεξέρχεται στις τροπολογίες 1 και 11. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, Θα ήθελα να πω ότι το να κάνουμε αγωγούς για φυσικό αέριο που να η προέλευση του είναι η Ρωσία δεν ξέρω κατά πόσο εξυπηρετεί το στόχο της ασφάλειας εφοδιασμού. Επανέρχομαι στις τροπολογίες του εισηγητή. Η παράταση του χρόνου που χρειάζεται για να καλύψουμε τις προδιαγραφές είναι κάτι το οποίο είναι λογικό σε ό,τι αφορά την κατασκευή νέων <clears throat> υποδομών, τροπολογίες 17 και 18. Υποστηρίζω επίσης τον εισηγητή σε ό,τι αφορά τη δημιουργία, την λειτουργία της ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο, που πρέπει να εμπλέκεται σε, όλες τις, σε όλα τα επίπεδα και να δίδει πληροφορίες στην Κομισιόν και σε προληπτικό επίπεδο και σε επίπεδο αντιμετώπισης κρίσεων, λόγω της εμπειρογνωμοσύνης των μελών της, αυτή η Επιτροπή θα πρέπει, αυτή η ομάδα θα πρέπει να θεωρείται ένα σημαντικό σώμα. Και νομίζω ότι ο εισηγητής δίνει σε αυτή την ομάδα ε, συντονισμού ευρύτερες εξουσίες από αυτές που προτείνει η Κομισιόν. Δεν αντιμετωπίζουμε σήμερα τον κανόνα του νήμιον 1, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η διαδικασία την οποία προβλέπει ο εισηγητής για να συζητήσουμε το θέμα αυτό και σε ποιο χρονικό ορίζοντα. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η χρήση του κανόνα νημιον 1 ή όχι. Εδώ θα πρέπει να θέσουμε και το θέμα της ε, ασυμβατότητος των κανόνων για υποδομές και για τους κανόνες τροφοδοσίες. Το ένα, το θέμα της τροφοδοσίας αφορά μονάχα προστατευμένους καταναλωτές, ενώ ο άλλος κανόνας του νήμιον 1 αφορά υποδομές οι οποίες έχουν γενικό χαρακτήρα χωρίς να υπάρχει υποχρέωση για την ασφάλεια τροφοδοσίας σε ίδιο επίπεδο σε όλα τα κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη μορφή συμβιβασμού του, της προδιαγραφής νήμιον 1 και των επενδυτικών αποφάσεων και ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κανόνας νήμιον 1 για την αξιολόγηση της επίτευξης ασφάλειας εφοδιασμού. Έχουμε ακούσει πολλές φορές τη συζήτηση αυτή ότι θα οδηγήσει σε μια στρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας και ένα απατηλό αίσθημα ασφάλειας στους καταναλωτές. Δεν επαρκεί λοιπόν η εφαρμογή του κανόνα νήμιον 1 γιατί αφήνει περιθώριο σε ευρύτητα ερμηνεών. Θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη ιδέα για τις επενδύσεις οι οποίες είναι απαραίτητες. Ίσως χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να διευκρινίσουμε καλύτερα τον ρόλο του κανόνα νήμιον 1 σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση κινδύνου γιατί θα πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε χώρα λαμβάνοντας υπόψη τις ε, ιδιαιτερότητε κάθε χώρα για να δικαιολογήσει τη δημιουργία περαιτέρω επενδύσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι πληροφορίε οι οποίε είναι από εμπορική άποψη, ε, εγώ θα καταθέσω και άλλε τροπολογίε πέραν αυτή του εισηγητή για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη εμπιστευτικότητα για τα δεδομένα τα οποία είναι στα χέρια των, των ρυθμιστικών αρχών και της Κομισιόν γιατί αυτό έχει επίπτωση στις επενδυτικές αποφάσεις θα θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η Κομισιόν και οι άλλοι ρυθμιστικοί φορείς εξασφαλίζουν απόλυτη εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Τέλος για το θέμα των προστατευμένων καταναλωτών. Θέλω να υπάρχει κάποια ευελιξία για τα κράτη-μέλη για να καθορίσουν αυτά τι θέλουν να <clears throat> περιλάβουν στον κατάλογο των προστατευμένων καταναλωτών. Αυτό που θέλουν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της χώρας τους. Και θα πρέπει όμως παράλληλα να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο για το ποιοι είναι αυτοί που θεωρούνται προστατευμένοι πελάτες σε κάθε χώρα μέλος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στοστόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει το πρόβλημα χρόνου το οποίο λαμβάνω υπόψη μου και γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομο, παρά το γεγονό ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα το οποίο είναι ε, πολύ πλοκό και πολύ ευρικό και το οποίο αξίζει μια ευρύτερη συζήτηση. Εγώ θέλω να εξάρω το έργο του κυρίου Βιδάλ Κουάδρα. και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η προβληματική που αντιμετωπίζει ο κύριος Βιδάλ Κουάδρα, ιδίω μετά την κρίση του προηγουμένου Γενάρη. Και είναι γεγονό ότι είναι μια πολύπλοκη προβληματική. Θα πρέπει να μην περιπλέξουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση στην αγορά φυσικού αερίου που λειτουργεί με περαιτέρω κανόνες και προδιαγραφές. Αλλά, όπως είπε και ο συγητής, είναι απαραίτητο να έχουμε κανόνες για την αντιμετώπιση κρίσεων <clears throat> ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις από ευρωπαϊκές αρχές και να μην αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό αποκλειστικά και μόνο σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό έχω να θέσω ένα ερώτημα για το, την παράγραφο 29 που αφορά ορισμένους μηχανισμούς που ενεργοποιούνται εάν υπάρξει μια απόκληση της τάξεως του 10% σε σχέση με την τροφοδεσία. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευαίσθητο. Μπορεί να καλύπτει ακόμα και μια ένα τεχνικό σφάλμα και μια ε, τροποποίηση της ροής σε επίπεδο μιας μέρας και μόνο. Θα είναι πολύ δάπανο να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα τεχνικά προβλήματα εάν δεν πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν πρέπει λοιπόν όταν είναι τόσο μικρό το κατόφλι να έχουμε ένα τόσο μικρό κατόφλι. Εγώ νομίζω πρέπει να θεσπίσουμε ένα κατόφλι της τάξης του 20% ή και παραπάνω. Γι' αυτό θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο σημείο αυτό ώστε να έχουμε ένα κατόφλιο το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα ένα ακόμα θέμα. Έχει αναφερθεί και το θέμα του υγροποιημένου φυσικού αερίου και της χρησιμοποίησής του και εγώ θα υποστήριζα να αναφερθούμε και, το, και στο φυσικό αέριο υποπίεση όπου είναι πιο εύκολη η μεταφορά του και δεν ε, περιέχει τεχνικά προβλήματα. Κυρία Χόλ, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει και τις λεπτομέρειες που μας παρουσίασε, διότι πραγματικά είναι ιδιαίτερα περίπλοκο να παρουσιάσουν, να υποβληθούν σαφείς κανόνες που θα λειτουργήσουν σε περίπτωση κρίσης και ε, χαίρομαι ότι είπε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μέτρα που στηρίζονται στην αγορά ακόμα και σε περίπτωση κρίσης. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν. Η πρόταση αυτή κυρίως αναφέρεται στα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Όμως ο εισηγητής προτείνει και κάτι για να καλύψει τα μακροπρόθεσμα προβλήματα. Π.χ. Ε, νέες διασυνοριακές δομές ε, και αναδιάρθρωση των δικτύων και φυσικού αερίου. Εάν όμως αναφερθούμε σε αυτά τα μακροπρόθεσμα μέτρα, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την, το τομέα της ζήτησης. Και υπάρχει ένα ιδιαίτερα ευπρόζεκτο project το οποίο υιοθετήθηκε για, την, για να βελτιώσουμε την ενεργειακή αποτελεσματικότητα του αερίου στην Ουκρανία ε, θα πρέπει να ε, λαμβάνουμε υπόψη μας ε, και την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις τρίτες χώρες που μπορούν να προμηθεύουν την Ευρώπη. Δηλαδή, ίσως θα μπορούσαμε και στην έκθεση αυτή να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τα μακροπρόθεσμα σχέδια. Κύριος Γκούρεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο για το θέμα αυτό γιατί ήδη έχουν διατυπωθεί πολλά ερωτήματα στο θέμα αυτό και τα οποία ερωτήματα θα είχα θέσει και εγώ. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του και να αναφερθώ σε τέσσερα σημεία. Καταρχήν, η, ανάγκη της, η έννοια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και το κατόφλιο του 10%. Συμφωνώ με αυτό το κατόφλιο και την έννοια αυτή. Και επίσης αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος ε, Τούρμες και ο κύριος ε, Βιδάλ Κουάδρας, ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την περιφερειακή διάσταση στα σχέδια αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων. Το δεύτερο ερώτημά μου λοιπόν αφορά την ε, δυνατότητα αμφιδρόμων ροών ή πλευρικών ροών. Ξέρω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία, αλλά δεν μπορούμε να το εξασφαλίσουμε παντού. Αυτή η τροποποίηση της κύριας ροή λοιπόν, θα πρέπει να μπορεί να παίξει ρόλο σε ορισμένε περιπτώσεις και σε ορισμένα σημεία κομβικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις και μόνο θα πρέπει να εξασφαλίσει κανείς κατά πόσο οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές είναι έτοιμες να επομιστούν το κόστος για την δημιουργία αμφιδρόμων ροών. Τώρα, οι προθεσμίες για την εκτέλεση των έργων υποδομής, που είναι εδώ πάρα πολύ αυστηρά καθορισμένες, εδώ θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε σαφείς κανόνες για τα προγράμματα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για να καταλήξουμε και στη, στα σχέδια για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σχέδια όπως αυτά που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή απόδοση, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά. Θα πρέπει να αποφύγουμε την περίπτωση μέσα στις νομικές ε, διατάξεις που θα εφαρμόσουμε να δημιουργήσουμε ένα πρόσθετο διοικητικό και γραφειοκρατικό άχθος στα κράτη-μέλη και συγχρόνως δεν θα πρέπει να έχουμε πρόσφατο, πρόσθετο βάρος για την αγορά και πιθανές τρευλώσει. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν κύριε Ισίτα. Η κυρία Νίμπλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη γιατί περνάει ο χρόνος. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Βιδαλ Κουάδρας για τη θαυμάσια έκθεσή του. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση είναι η κατάλληλη για να αντιμετωπίσει την πρόταση της Κομισιόν, την πρόταση κανονισμού σε και να τη βελτιώσει σε διάφορα σημεία. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι λαμβάνεται υπόψη και ο ρόλος των επιχειρήσεων και βάσει των προτάσεων του εισηγητή μας εμπλέκονται πλήρως οι επιχειρήσεις και επίσης είναι σημαντικό ότι η ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο αποκτά κάποιες ε, αρμοδιότητες, έστω και τις διαφοροποιεί ο εισηγητής, έναντι της πρότασης της Κομισιόν. Επίσης, για τον κανονισμό της αμφίδρομης ροής. Το ερώτημα είναι πότε θα πρέπει να είναι υποχρεωτική αυτή η αμφίδρομη ροή. Είναι απαραίτητο να το περιορίσουμε λιγάκι σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Θέλω λοιπόν και πάλι να συγχαρώ τον εισηγητή για όλα αυτά τα στοιχεία. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι χρήσιμο να μπορέσει να υπάρξει και μια συζήτηση στην Επιτροπή μας σε κάποια χρονική στιγμή σε σχέση με τον κανόνα του νημιών 1 εγώ δεν έχω καταλήξει σε κάποια θέση με τον κανόνα του νη 1. Μα είχε πει ο αρμόδιο Γενικό Διευθυντή ότι δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστεί αυτό ο κανόνα, αλλά θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα να έχουμε μια πιο εντατική συζήτηση ακριβώ για το θέμα αυτό και το ίδιο ισχύει και με τον ε, ορισμό των προστατευμένων πελατών που με οδηγεί σε ορισμένε αμφιβολίε. Θα ήθελα εδώ να επανέλθω σε αυτό που είπε και ο κύριος Τοζενόσκι, έχω κάποιες αμφιβολίες κατά πόσο το κατόφλιο του 10% δηλαδή το πότε έχουμε μια συνολική κατάσταση έκτακτη ανάγκης, μήπως το κατόφλι του 10% είναι πολύ χαμηλό. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε τις απόψεις του, της Κομισιόν για το θέμα αυτό, να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα στην περίπτωση αυτή, γιατί πιστεύω ότι με το 10% σαν κατόφλι μπορούμε να έχουμε τον κίνδυνο να έχουμε μια υπερβολική αντίδραση σε μικρά προβλήματα. Ίσως το 20% θα είναι πιο πρόσφορο κατόφλι και γι' αυτό το ερώτημά μου θα ήταν ποια είναι η εμπειρία που έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμή και αν αυτή θα δικαιολογούσε να χρησιμοποιήσουμε ένα υψηλότερο κατόφλι. Ευχαριστώ. Σύμφωνοι. Η κυρία Παράσκα Μπομπίνσκα έχει το λόγο. σήμερα συζητούμε γενικές και μακροπρόθεσμα, γενικά και μικροπρόθεσμα προβλήματα, αλλά και κάποια πιο συγκεκριμένα η ασφάλεια του εφοδιασμού όπως είπε και Βαρόνια Άστον είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε στήσουμε σε κάποια, κάποια στιγμή σε κάποια συνεδρίαση αυτά τα θέματα γενικότερα και σε σχέση με την εξωτερική πολιτική να φτιάξουμε μια τέτοια ομάδα ούτως ώστε να μπορούμε να τα συζητήσουμε από κοινού τα θέματα αυτά στην οποία να είναι παρόντες όλοι οι συναρμόδιοι για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κάρετ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βινταλ Κουάντρας για την έκθεσή του που είναι βελτίωση, συνιστά βελτίωση σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέει ο Βιντάλ Κουάντρας για τη σημασία των μηχανισμών της αγοράς, ιδιαίτερα σε στιγμές κρίσης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να καταλάβουμε κιόλας ότι στην Ευρώπη, στα διάφορα μέρη της Ευρώπης, οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Η Κομισιόν αυτά που προτείνει ε, φαίνεται να αρμόζουν στην νοτιοανατολική Ευρώπη που, έχουν, ε, που έχει διασυνδέσεις ε, που και μπορούν να αντιμετωπίσουν μια κάποια διακοπή του εφοδιασμού αλλά στη Βόρεια Ευρώπη, στις τρεις βαλτικές χώρες και στη Φινλανδία είμαστε πλήρως απομονωμένοι από την υπόλοιπη Ευρώπη εμείς και υπάρχει μόνο μία σύνδεση με τη Ρωσία ο κύριος Τούρμες είπε ότι οι βαλτικές χώρες πρέπει να ε, συνεργάζονται μεταξύ τους. Ε, Του απαντώ ότι βεβαίως υπάρχει στενή συνεργασία. Αλλά νομίζω το 2005-2006 όταν ο χειμώνας ήταν ιδιαίτερα κακός ε, έγινε προσπάθεια να ε, διοχετευθεί αέριο σε όλους υπάρχει στις, βαλτικές χώρες υπάρχει στενή συνεργασία το θέμα δεν είναι συνεργασία εντός της Ευρώπης το θέμα είναι ότι η περιφέρεια αυτή η περιοχή για την οποία μιλώ έχουν μία μόνο διασύνδεση έναν μόνο αγωγό με τη Ρωσία όταν παραδείγματο χάνει πρέπει να γίνουν επισκευέ σε αυτόν τον αγωγό υπάρχει αμέσω πρόβλημα και εκεί πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση κοινοτικό επίπεδο. Το θέμα λοιπόν είναι πώς να δημιουργήσουμε μια αγορά δημιουργώντας διασύνδεση. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος τώρα θα πρέπει να επιταχύνουμε λίγο για να κλείσουμε δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά στον εισηγητή ο κύριος Χιλμπρέχτ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Βιντάλ Κουάδρας που παρουσίασε μια έκθεση η οποία ουσιαστικά διευκολύνει και εμένα το έργο μου εμπολής. Συμφωνούμε με τα σχόλια που κάνει ο εισηγητής και με κάποια άλλα σχόλια που έγιναν από του Σκιώδη Συγητή και άλλους συναδέλφους εδώ στην Επιτροπή ε, ιδιαίτερα σχετικά με το ρόλο της αγοράς και των ε, εταιριών και τις αντίστροφες ροές συμφωνούμε με όλα αυτά συμφωνούμε επίσης και ότι μέτρα που δεν βασίζονται στην αγορά θα πρέπει να παίρνονται μόνο σαν ε, τελευταία λύση αν δεν υπάρχει τίποτε άλλο θα ήθελα όμως ε, ε, θα ήθελα να αναφέρω τώρα πέντε θέματα ε, 15 για τις τροπολογίες 15, 16 και 51 θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια πρώτα πρώτα αυτό που ζητεί ο εισηγητής να υπάρχει σχέδιο επίγουσας κατάστασης σε κοινότικο επίπεδο δεν θα πρέπει να ε, είναι ε, το σχέδιο σχέδια αυτά να επιβάλλονται άνωθεν αλλά θα πρέπει να ξεκινούν από τη βάση η Κομισιόν θα πρέπει απλώς να συνθέτει ορισμένα πράγματα και να τα και να τα εφαρμόζει δεν μπορεί να επιβάλλονται άνωθεν ορισμένα πράγματα Επίσης, ορισμένα πράγματα μπορούν να γίνουν μόνο όταν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία. Ο κ. Τούρμες είπε ότι η Κομισιόν πρέπει να παίρνει ορισμένα στοιχεία συγκεντρωμένα με ένα συγκεκριμένο τρόπο κτλ. Ωραία, αυτό είναι γεγονό. Απ' την άλλη μεριά ζητάτε να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ορισμένα πράγματα. Αυτά είναι λίγο αντιφατικά εάν η Κομισιόν δεν έχει τα στοιχεία τα οποία μπορεί να επεξεργαστεί. Δεύτερο σχόλιο για τις τροπολογίες 12 και 17 παρά για τις ε, προθεσμίες ο εισηγητής ε, μιλάει για τρία με πέντε χρόνια παράταση εμείς πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό αναγνωρίζουμε τον επίγοντα χαρακτήρα των μέτρων και πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε τα κράτη-μέλη όμως ε, κάποιες ε, ε, αντιμετωπίσεις ε, τύπου επενδύσεων παραδείγματο χάρη χρειάζονται παραπάνω χρόνο ίσως έχει δίκιο ο κύριος Σφόμποντα που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενδιάμεση έκθεση μετά από τρία χρόνια για να δούμε τι έγινε και τι δεν έγινε πριν προχωρήσουμε τρίτο θέμα που θα ήθελα να θέσω σχετικά με τροπολογία 24 αν κατάλαβα καλά θέλει ο εισηγητής να διαγράψουμε μια παραπομπή που μια αναφ... μάλλον να κάνουμε μια αναφορά στις εμπορικές συμβάσεις που αναφέρονται ε, εμείς νομίζουμε ότι το κείμενο είναι καλό σε συγκεκριμένη περίπτωση επίσης να πω μερικά πράγματα για το συντονισμό ξέρω ότι για πολλούς και για τον εισηγητή ο συντονισμός είναι πολύ σημαντικό εργαλείο αλλά καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι υπαρβάλλουν ορισμένοι συνάδελφοι σε αυτά που λένε γιατί αυτή η ομάδα συντονισμού δεν είναι αρχή δεν είναι σαν τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών δεν είναι αρχή θεσμικό όργανο σαν την Κομισιόν άρα δεν μπορούμε να δώσουμε δικαιώματα και εξουσίες στην ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο ε, πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο το οποίο πρέπει να εμπλέκεται αλλά παραμένει συμβουλευτικό όργανο η Κομισιόν θα πρέπει να δρά δεν μπορούμε να πούμε ότι το, ο, η Κομισιόν πρέπει να περνάει πάντα από αυτή την ομάδα ή ότι η ομάδα αυτή έχει κάποια προνόμια. Αυτό είναι υπερβολικό κατά την άποψή μου. Το πέμπτο θέμα που θα ήθελα να σχετίζεται με τροπολογία 29 ελέγχθη ότι η έκτακτη ανάγκη κηρύσσεται μόνο αν άνω της μιας ρυθμιστικής αρχής κηρύξουν έκτακτη ανάγκη. Μα θα πρέπει να είμαστε λίγο συνεπείς νομίζω ότι μπορούμε να επιτρέψουμε ακόμη και μία ρυθμιστική αρχή να ζητήσει να γίνουν ορισμένα πράγματα αν υπάρχει ανάγκη. Τώρα η κυρία Νίμπλε αλλά και ο κύριος Στοζενόφσκι είπαν ότι το κατόφλι του 10% είναι υπερβολικά χαμηλό. 10% εισαγωγών από τρίτες χώρες μιλούμε εδώ, λέμε εδώ και οι εισαγωγές θα αυξηθούν δηλαδή 10% είναι αρκετά σημαντικό ποσοστό και βεβαίως δεν θέλουμε να υπάρχουν αυτοματισμοί αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας να μπορεί να εκτιμήσει η Κομισιόν κατά πόσο 10% είναι σημαντικό για κάποια περιφέρεια ή για, κα... για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ νομίζω ότι το 10% είναι το σωστό επίπεδο, 20% είναι υπερβολικά ψηλό, το είδαμε αυτό στο παρελθόν. 20% κατόφλι σημαίνει ότι θα ξεσηκωθεί όλη η Ευρώπη όπως είδαμε και με την τελευταία κρίση γι' αυτό μιλάμε για 10% εδώ να κάνω και μερικά σχόλια τώρα για μερικές από τις παρατηρήσεις που έκαναν οι άλλοι συνάδελφοι Βεβαίω θέλουμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή για τα δύο κρεμούντα θέματα, το 1-1 και τους προστατευμένου πελάτε Από τεχνική απόψεως πρόκειται για πολύ δύσκολα θέματα, είναι δύσκολο να βρεθούν συμβαστικέ λύσει. Συνεργαζόμαστε επίση και με τη βιομηχανία και ελπίζουμε να βρούμε ε, τον τεχνικά σωστό ορισμό του 1-1 αλλά μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε αυτά και με τον κύριο Βιντάλ Κουάντρα ώστε να μπει στη τελική έκθεση ο νέο ορισμό. Τώρα οι προστατευμένοι πελάτες είδαμε ότι υπάρχουν ε, και διεστάμενες απόψει απόψεις εδώ στην Επιτροπή ίσως λοιπόν πρέπει να το αναθέσουμε το θέμα στα κράτη-μέλη να βάση την αρχή της επικουρικότητας λένε, ορισμένοι άλλοι λένε ότι ίσως πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εναρμόνιση για να μην υπάρχει διαστρέβλωση της ροής του αερίου με τα, στα κράτη-μέλη. Ίσως θα πρέπει να βρούμε μια κάποια λύση στη μέση, να υπάρχει ένας ορισμός αλλά να υπάρχει μια διακριτική ευχέρια για τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό πρέπει να το συζητήσουμε και με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο και μετά βεβαίω θα έρθουμε σε επαφή με τον εισηγητή για να βρούμε τον τελικό ορισμό ο οποίος να ικανοποιεί και τους μεν και τους δε και αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να λειτουργήσει η εσωτερική η ενιαία αγορά και του εκείνους που πιστεύουν ότι κάποιες ιδιαιτερότητες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Έγινε και μια άλλη παρατήρηση για την κατάσταση της Βαλτικής, της περιοχής της Βαλτικής, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Κάλεντ και ο κ. Σολτάρκας αναφέρθηκαν στα θέματα αυτά και είπαν ότι χρειάζονται νέες διασυνδέσεις. Ευχαριστώ την προσοχή σας στο έργο του Μπέμιτ. Ε, υπάρχει αυτή η υψηλού επίπεδου ομάδα για τα θέματα αυτά των διασυνδέσεων. Κάναμε πρόοδο στα θέματα της ηλεκτρικής ενέργειας, στο Βίλνεος, ε, κατά, είδαμε, ε, ότι υπάρχει μεγάλη, πολύ καλή συνεργασία αλλά βεβαίως ακόμη περισσότερα μπορούν να γίνουν για το φυσικό αέριο οι αποθήκες της Λετωνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω περαι, περισσότερες ε, διασυνδέσεις με τη Δύση, με το Βορρά, με την Νορβηγία αυτά είναι όλα εφικτά και υπάρχει και ο αγωγός από την Νορβηγία στη Βαλτική, στην Πολωνία αυτό το σχέδιο βέβαια προς το παρόν καταργήθηκε και αναβλήθηκε ε, πρέπει να τα ξαναδούμε όμως όλα αυτά και το, η ομάδα που δημιουργήθηκε είναι χρήσιμο εργαλείο νομίζω θα τα δούμε αυτά και στο μέλλον η κυρία Βαλεάν μίλησε για το στάνταρ N-1 είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ε, δεσμευτική σχέση μεταξύ αυτού του στάνταρ και των επενδύσεων σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει τέτοια σχέση και όπως δικαίως είπατε η, το N 1 ένα θα πρέπει να σχετίζει, να βασίζεται αν θέλετε στην απόφαση της, στην κρίση της αρχής της αρμόδιας αυτό είναι κομμάτι της όλης ε, η φιλοσοφίας του 1-1 αυτά κύριε πρόεδρε προσπάθησα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που έγιναν ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Υπάρχουν προφανώ διστάμενε απόψει μεταξύ του Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, όπως ξέρουμε και από το παρελθόν. Κύριε Βιντάλ θέλετε να προσθέσετε κάτι. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπήρχε εδώ διατύπωση της επιθυμίας να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Μετά από αυτά που άκουσα από τους συναδέλφους, αν μόνο εμείς έπρεπε να φτάσουμε μια συμφωνία, προφανώς θα είχαμε φτάσει σε μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, γιατί υπάρχει ευρεία συνένεση. Δυστυχώς δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε από την απέναντι πλευρά το Συμβούλιο. Και είναι γενικό, γενικά μεγάλο το επίπεδο συνένεση που βρίσκουμε στην Επιτροπή μας, αλλά φοβάμαι ότι δεν βρισκόμαστε στο διομικό σχήματος απόλυτα με το Συμβούλιο. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια συμφωνία σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης αλλά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό τελικό αποτέλεσμα. Για τις παρατηρήσεις που διατυπώσαν οι συνάδελφοι και που εκφράζουν την ε, συμφωνία τους με την έκθεσή μου ή να διαφοροποιηθούν σε ορισμένα σημεία αλλά ακολουθώντας την οδική, ε, το οδηγό νήμα της έκθεσής μου εγώ δεν θα αναφερθώ γιατί θα είναι επαναληπτικό να κάνω κάτι τέτοιο. Υπάρχουν κάποια σημεία για τα οποία θέλω να κάνω ορισμένε διευκρινήσει. Όταν μιλάμε για το κοινωνικό, κοινοτικό συγγνώμη, σχέδιο δράση, δεν μιλάμε για να υπάρξει ακόμα ένα επιπλέον σχέδιο, όχι μιλάμε για να υπάρξει κάποια καλύτερη εναρμόνιση και παρακολούθηση των εθνικών σχεδίων. Δεν μιλάμε για ένα επιπρόσθετο ε, σχέδιο Τη Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε για την επίτευξη συνεκτικότητα μεταξύ των εθνικών σχεδίων, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούν να είναι και αποτελεσματικά. Για το θέμα των τριών ή πέντε ετών. Νομίζω ότι η πρόταση του κ. Σφόμποντα μας δίνει τη σωστή αντιμετώπιση. Ένα ενδιάμεσο στάδιο δηλαδή και μετά ανάλογα με την πρόοδο να προχωρήσουμε <clears throat> βάσει μιας ενδιάμεσης Αξιολόγηση σε ενδεχόμενη παράταση για δύο χρόνια. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Όταν διαγράψαμε <clears throat> τις εμπορικές συμφωνίες, αυτό έγινε σε ένα άρθρο γιατί αναφέρονται σε άλλα άρθρα. Οι μηχανισμοί αντιστάθμισης και αποζημίωσης προφανώς θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο κανονισμό, αλλά μόνο στην περίπτωση θεμάτων που δεν καλύπτονται από τους, μηχανικούς, από τους μηχανισμούς της αγοράς. Έχει νόημα αυτό. Για το ρόλο της ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο, προφανώς η ομάδα αυτή δεν είναι μια αρχή, αυτό είναι προφανές, αλλά ούτε μπορεί να είναι ένας βουβός μάρτυρας των τεκτενομένων. Η ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο έχει κάποιο ρόλο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε, να εξειδικεύσουμε το ρόλο του και να τροποποιήσουμε τη διατύπωση για να μην υπάρχουν αμφισημίες. Αλλά Νομίζω ότι συμφωνούμε μεταξύ μας ότι αυτή η ομάδα συντονισμού έχει κάποιο προεξάρχοντα ρόλο, λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό φυσικά ότι δεν έχει αποφασιστικό ρόλο, δεν είναι μια αρχή για τα θέματα αυτά. Συμφωνούμε λοιπόν εκεί. Αν σα φαίνεται αμφίσιμη η διατύπωση, μπορούμε να την τροποποιήσουμε και να την βελτιώσουμε. Επίση, θέλω να αναφερθώ σε ένα σημείο το οποίο έθεξε ο κ. Γκάιτ. Είναι γεγονό ότι οι βαλτικέ χώρε έχουν μια διαφορετική ιδιαιτερότητα. Είναι μια χωριστή περίπτωση διαφορετική η προβληματική τους από την Ανατολική Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, το κατανοούμε αυτό. Αλλά όταν εμείς θέλουμε να θεσπίσουμε προτεραιότητες για τις επενδύσεις, προφανώς θα λάβουμε υπόψη ιδιαίτερη, ιδιαίτερα την περιοχή της Βαλτικής και τη διασύνδεσή της με την υπόλοιπη Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και είναι προτεραιότητα η διασύνδεση των χωρών της Βαλτικής μέσα στο πλαίσιο αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το θέμα αυτό η ανησυχία επίση της κυρίας Χολ για την εισαγωγή αυτών των, σε αυτά τα σχέδια μέτρων ζήτηση, δηλαδή εξέβρεσης ενεργειακής απόδοσης, προφανώς δεν έχω καμία επιφύλαξη για αυτό το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, μετά από όλα αυτά που άκουσα, νομίζω ότι είναι πολύ καλή η θέση μας. Και η κυρία Βομπίνσκα είπε κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ορθό και σόφρον. Ότι λόγω της γεωπολιτικής διάστασης του θεμάτος αυτού είναι απαραίτητη και καλύτερη επίτευξη συντονισμού μεταξύ της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενεργειακής πολιτικής. Δηλαδή η ιδέα να ακούσουμε την άποψη από κοινού της κυρίας Άστον και του νέου Γερμανού Επιτρόπου του κ. Έτσιγκερ, που είναι αρμόδιος για την ενέργεια νομίζω ότι είναι μια πολύ θετική ιδέα. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος αυτού, μια καλύτερη ανατένιση, γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι χωρίς την γεωπολιτική διάστασή του αυτό το θέμα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στην πληρότητά του. Αυτά λοιπόν κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ λέει και ο Πρόεδρος. 14 Ιανουαρίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Έχουμε, μία, έχουμε μισή ώρα μόνο και τρεις, τρία θέματα να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ να επιταχύνουμε λιγάκι την εργασία μας και ζητώ από την κυρία Τρότμαν να μας ε, αναφέρει τα, ε, να μας κάνει μια έκθεση για την, έκθεση, για την συνάντηση, μάλλον για τη διακυβέρνηση του ίντερνετ στο Σάμα Σέιχ. Έχετε το λόγο κυρία Τρότμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ξέρω ότι είναι μετρημένος ο χρόνος μας και θα ήθελα να τα μοιραστώ αυτά τα οποία έγιναν και με τα μέλη της Επιτροπής μας. Συμμετείχαμε στο τέταρτο φόρουμ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου Είμαστε μια αντιπροσωπεία από την οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από τέσσερις επιτροπές, από την ΣΤΟΑ, από την Επιτροπή πολιτισμού. Η κυρία Καστίγιο, η οποία θα έπρεπε να ήταν μέλος της αντιπροσωπείας μας, τελικά δεν μπόρεσε. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστήσεις τις ευχαριστίες μου στον κύριο Μαρτίνο Σά, ο οποίος είναι υπεύθυνο των υπηρεσιών της Επιτροπής μας, διότι με την αντιπροσωπεία του κύριου Νίμπελ, του κύριου Φόρτη και των δύο φυλάκων αγγέλων μας κατάφεραν να ασχοληθούμε με τα σημεία της ημερήσιας διάταξης, τα οποία ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητα. Να μιλήσω γι' αυτό το, τα χαρακτηριστικά του τέταρτου Φόρουμ και του, του απολογισμού που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Διαπιστώσαμε πόσο αλλάξαν τα πράγματα από την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε στην Αθήνα, στο πρώτο φόρουμ διακυβέρνηση του διαδικτύου. Για το βασικό θέμα που αφορούσαν την συνέχεια, τη συνέχιση της διακυβέρνησης ε, του διαδικτύου και διευκρινίζω για τους συναδέλφους που δεν γνωρίζουν το σύστημα αυτό των διεθνών συναντήσεων που δεν αποτελεί έναν επίσημο οργανισμό που, από, που παίρνει παίρνει αποφάσεις, αλλά είναι μια πλατφόρμα συζήτησης, ένα βήμα συζήτησης για θέματα συγκεκριμένα, τα οποία αφορούν όλους μας, μέσα σε μια τεχνική πολυσυμμετοχική, αν θέλετε. Εμείς οι Ευρωπαίοι μιλήσαν ε, με μια φωνή, η Σουηδική Προεδρία, η κυρία Ρέντινγκ, η Επίτροπος και εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητήσαμε να, υπάρξει, να δοθεί συνέχεια στη διακυβέρνηση του διαδικτύου στο EGF, ότι θεωρούμε ότι δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις με τον τρόπο αυτό να βρεθούν λύσεις σε διάφορα τεχνικά και τεχνολογικά προβλήματα, να εξετάσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες το τι σημαίνει δημόσια υπηρεσία, η υπηρεσία μέσω ίντερνετ, ποια είναι τα δικαιώματα του κοινού, ποια είναι η θέση των κυβερνήσεων, ποια είναι η θέση του κράτους, ποια είναι η θέση των χρηστών και με τον τρόπο αυτό μπορούμε ναι από το διεθνές επίπεδο να περάσουμε από το εθνικό επίπεδο και να φτάσουμε σε επίπεδο χρήστη, ατομικού χρήστη του διαδικτύου. Επομένως θεωρούμε ότι υπάρχει ε, μια θετική εξέλιξη ε, μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα βέβαια αλλά τέλος πάντων θα μπορούσαμε ε, και να στραφούμε και προς τις αναδυόμενες χώρες και στις χώρες που ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικές η Κίνα ας πούμε οι χώρες αυτές οι επιφυλακτικές δεν βρίσκονται σε ένα τέλειο επίπεδο δημοκρατίας και να το, για να μιλήσω και έτσι και διπλωματικά. Ορισμένες ε, χώρες ε, είναι έτοιμες να ε, δεχτούν το τέλος ε, της ε, διακυβέρνησης του, του διαδικτύου και να μετατραπεί αυτό το φόρουμ σε μια διακυβερνητική συνεργασία, δηλαδή να έχουμε ένα δεύτερο ΟΗΕ, το οποίο σημαίνει βέβαια και μια αποδυνάμωση για να μην πω και μια κατάργηση της συμμετοχής της, ε, του, του, της κοινωνίας των πολιτών. Δεύτερο θέμα πάνω στο οποίο συζητήθηκε και έντονα συζητήθηκε ήταν η μεταμόρφωση του ICANN, η, η ανεξαρτησία από το Υπουργείο Εμπορίου των, των Ηνωμένων Πολιτειών για, και να δούμε πώς θα καθοριστεί η ε, ε, καθορίζεται από την νομοθεσία της, ε, της Καλιφόρνιας θα γίνεται κάτι άλλο ε, θα γίνει πιο διεθνές δηλαδή ακούστηκε και η Γενέβη δηλαδή ένας χώρος ο οποίος είναι πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έστω και αν δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθεαυτή ένα άλλο σημείο το οποίο ε, συζητήθηκε και με τις αντιπροσωπείες που συναντήσαμε αλλά και με τον πρόεδρο της ICAN είναι το θέμα των reviews, των αναθεωρήσεων δηλαδή της ε, εξέλιξης ε, της Επιτροπής αυτής του ίντερνετ για την απονομή των ονομάτων και των αριθμών. Συζητήσαμε με τον κύριο Γιάννη Σκάτλινγκς ο οποίος είναι ο πρέσβης της Λετωνίας της Εστονίας στην Γαλλία. Διαπιστώσαμε κάποια σημεία που ε, προσθέτουν αν θέλετε έναν ε, επιπλέον χαρακτήρα, ενδυναμώνει τον χαρακτήρα μας, παραδείγματο χάρη η προστασία των παιδιών, ε, κάτι το οποίο εμείς συζητήσαμε, είναι πολύ σημαντικό για μας και θεωρούμε ότι έχουμε ενδυναμώσει το σύστημα. Δεύτερον είναι για τα ονόματα των διαφόρων τομέων, τα generic ε, topic domains. Αυτό είναι ένα θέμα ε, για το οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Είναι θέματα δηλαδή που έχουν παραμείνει σε εκκρεμότητα, είναι ανοιχτά και πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω. Ε, τα critical resources τώρα έγινε μια συζήτηση που θα πρέπει να συνεχιστεί για τα INA. Θα πρέπει να συζητήσουμε και τα θέματα προσβασιμότητας, τα θέματα ασφάλειας και τα προβλήματα διακυβέρνησης αυτής καθεαυτής. Έχουμε Έχουμε δηλαδή ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις, κάποιες συζητήσεις που πρέπει να εμβαθύνουμε και ε, που θα πρέπει να επαναληφθούν, κυρίως όσον αφορά την διακυβέρνηση, όχι μόνο και για το ICAN αλλά και για το ITU. Ε, μπλεχτήκαμε αν θέλετε άμεσα με, την, ε, με τις δύο αυτές επιτροπές ICAN και IU για, για να δούμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες οι αυτών των δύο οργανισμών και η θέση μας είπαμε ότι η ITU είναι υπεύθυνη και αρμόδια για τα θέματα υποδομών και η ICAN θα αναλάβει την ε, διαχείριση των ονομάτων και των πτυχών του ίντερνετ. Αυτή ήταν μια θέση η οποία εκτιμήθηκε και θετικά κιόλα. Επίσης του χρόνου είπαμε ότι μέσα στα πλαίσια τη προετοιμασία του πέμπτου φόρουμ ε, στην Λιθουανία αυτή τη φορά θα έχουμε μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή παρουσία η οποία την και ευθύνη ε, θα η Λιθουανία, η Ισπανική Προεδρία και η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίξουν με ένα μείζωνα ρόλο. Η προετοιμασία αυτή βέβαια πρέπει να ξεκινήσει γρήγορα, διότι η συνάντηση ε, στη Λιθουανία θα γίνει το Σεπτέμβρη και όχι τον Νοέμβριο όπως συνήθως συναντιόμαστε. Ε, δεύτερον, θα ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πολιτικά θέματα, τα δύσκολα πολιτικά θέματα, αλλά και την προετοιμασία του νέα, της νέας φάσης, του νέου σταδίου, εάν είμαστε έτοιμοι βέβαια. Γι' αυτό ξεκινήσαμε συζητήσεις με μια αντιπροσωπεία της α, ε, νότιας της Σαχάρας Αφρικής, διότι η Κένια μετά την Λιθουανία θέλει να υποδεχθεί την... Ε, το επόμενο φόρουμ του, του, της που θα είναι το βελτιωμένο ε, ε, ΙΖΕΦ, γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά μαζί του. Πώ μπορούμε να προετοιμάσουμε όλα αυτά. Καταρχάς να έχουμε μια συνάντηση με του εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, όπω είπαμε και με τη Γαλλίδα Υπουργό, να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία μετά την συνάντηση του Σάρμελ Σίκ ε, και μέσα στα πλαίσια τη Ένωση για τη Μεσόγειο και μετά ε, να ε, συναντήσουμε και να συζητήσουμε και με τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ ε, για το που είναι υπεύθυνο για το ΙΖΕΕΦ και να συζητήσουμε τα θέματα της Κένιας και της νότιας της Σαχάρας Αφρικής. Επίσης συζητήσαμε και με την αντιπροσωπεία της Βραζιλίας πέραν των Αφρικανικών. Είχαμε μια συνάντηση με τον Υπουργό Τελεπικοινωνιών της Αιγύπτου, μια συνάντηση με την αντιπροσωπεία που, της Ινδίας που θέλει να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί μας, μια συνάντηση με την Εθνική Αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου αποφασίσαμε κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία, στα οποία αναφέρθηκα και εκείνοι θέλουν να συνεργαστούν στενά μαζί μας. Συναντήσαμε το Συμβούλιο της Ευρώπης, μια συνάντηση με την ICAN, την ITU, μια συνάντηση με την Σουηδική Προεδρία και τους εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών. Αυτά. Πρόεδρε. Είδατε ότι δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά, πέραν των διάφορων, των διαφόρων workshops, ε, μπορέσαμε να συμμετάσχουμε, να συζητήσουμε, να ενημερώσουμε τους συνομιλητές μας για, το, ε, για τα επόμενα προγράμματα, για την επόμενη χρονιά, το ΣΠΕΚΤΡΑ, τα, τις ηλεκτρονικές πολιτικές, ε, τις οικουμενικές υπηρεσίες και τον ρόλο μας ε, στην διατήρηση του φόρμου διακυβέρνησης του διαδικτύου. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν δεν βιαστούμε δεν θα μπορέσουμε να τελειώσουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν να είσαστε λακωνικοί. Δύο ομιλητές, αν μπορείτε να περιοριστείτε σε ένα λεπτό, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να προλάβουμε τα άλλα θέματα. Κυρία Κοχμερίν, ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω και την κυρία Τροτμάν φυσικά για την έκθεσή της Χθε έγινε και η ετήσια ομιλία της ΣΤΟΑ για ένα διαδίκτυο το οποίο θα είναι ανοιχτό σε όλους και ήταν πολλοί συνάδελφοι από την Επιτροπή μας παρόντες θέλω να τους ευχαριστήσω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προφανώς έχει να αναλάβει ένα ιδιαίτερο ρόλο σε σχέση με αυτή την προβληματική της πρόσβασης στο ίντερνετ που θεωρούμε ότι είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών και γι' αυτό η σημαντική συμμετοχή μας και στα διεθνή φόρα και θέλω να τονίσω ότι και αυτό θα πρέπει να είναι από τα βασικά σημεία στην ακρόαση τη αρμόδια επιτροπού, γιατί δεν είναι μονάχα ένα τεχνικό θέμα, αλλά είναι ένα πραγματικό θεμελιώδη δικαίωμα για όλου του πολίτε τη Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στρακατέλη. Έχετε το λόγο. Ένα λεπτό. Θα συμφωνήσω με την προηγουμένη ομιλήτρια το ζήτημα του ίντερνετ είναι ένα ζήτημα που έχει ε, θεμελιώδη ε, κοινωνική σημασία, πρακτικώς μεταβάλλει όλους τους τρόπους ε, δημοκρατικής διακυβέρνησης ή παραγωγικών διαδικασιών. Θα ήμουν ευτυχής εάν το, η Επιτροπή μας και ίσως η ΣΤΟΑ αναλάμβανε μια δραστηριότητα σχετικά με την μελέτη των ζητημάτων που σχετίζονται με το ίντερνετ και δεν έχουν να κάνουν μόνο με την τυπική διάρθρωση λειτουργίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ζητώ την κατανόησή σας και σας ζητώ συγγνώμη που σας ε, ανέφερα ως κύριο Τσακατέλη. Πάμε στο σημείο 7, καταπολέμηση του καρκίνου. Η κυρία Γκροστέτη έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και θα το αντιμετωπίσουμε σε ένα τέταρτο. Είναι σημαντικό γιατί στην αίθουσα αυτή υπάρχει το 1 τρίτο των ατόμων που θα ε, το απασχολήσει το θέμα αυτό. Διότι ένα άτομα στα τρία κάποια στιγμή στη ζωή του στην Ευρώπη θα παρουσιάσει έναν καρκίνο. Δηλαδή 3,2 εκατομμύρια άτομα. Ξέρετε ότι η κατανομή του καρκίνου δεν είναι ισότιμη στην Ευρώπη και ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Υπάρχει ένα πραγματικό πρόγραμμα, γι αυτό, πρόβλημα, συγγνώμη, γι' αυτό και η Κομισιό μας κάνει μια πρόταση να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή συνεργασία όπου θα συμμετέχουν όλοι οι οργανισμοί για την καταπολέμηση του καρκίνου, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα, ένα ευρετήριο, αν θέλετε, των κενών, των προβλημάτων που υπάρχουν, να δούμε πώς μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις διάφορες ανάγκες και αυτή η συνεργασία κατά τη διάρκεια της περίοδου 2009-2013 έχει σαν στόχο να καταπολεμήσει, να βοηθήσει τις χώρες να καταπολεμήσουν τον καρκίνο, ε, δημιουργώντας ένα πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει την απογραφή, την ανταλλαγή πληροφοριών, ε, να δούμε ποιες είναι οι ικανότητες, ποιες είναι οι αρμοδιότητες, να αφορά την πρόληψη της ε, ασθένειας, αλλά και την καταπολέμηση της ασθένειας. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία αναφέρονται σε αυτή την ανακοίνωση. Καταρχάς η πρόθεση τη υγεία, η έγκαιρη ανείχνευση του καρκίνου, διότι το 1 τρίτο των καρκίνων είναι προβλέψιμοι και μπορούμε να του προλάβουμε, γιατί η πρόληψη αποτελεί την πιο, την πιο αποτελεσματική και οικονομική μακροπρόθεσμα ε, στρατηγική για την καταπολέμηση του καρκίνου. Η συνεργασία αυτή θα έχει σαν στόχο να δημιουργήσει δομέ παρέμβαση έτσι ώστε να έχουμε έναν τρόπο ζωή σε πιο υγιή να έχουμε μία έγκαιρη πρόληψη της ε, ε, ασθένειας, κυρίως αναφορά αφορά την ε, πρόληψη του καρκίνου του στήθους, του παχαίου σεντέρου, του τραχύλου της μήτρας, να μπορέσουμε να περιορίσουμε τα ποσοστά για του καρκίνους αυτού, διότι γίνεται αυτό. Δυστυχώ δεν έχουμε φτάσει στου αριθμού που θέλουμε. Επίση, θα πρέπει οι εξετάσει ε, να καλύψουν το 100% του πληθυσμού, διότι αν γίνει αυτό θα εξαφανιστεί, θα εξαλειφθεί ο καρκίνο αυτό. Ε, δεύτερον, διάδοση καλών πρακτικών ε, υγιεινή και που συνδέονται με τον καρκίνο. Αυτέ οι καλέ πρακτικέ θα μα επιτρέψουν να ευνοήσουμε την χρησιμοποίηση ομάδων όπου θα συμμετέχουν πολλέ ειδικότητε ε, και θα έχουν ε, όλα αυτά σαν στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής και για τους ασθενείς. Ξέρουμε ότι οι ανισότητες είναι τεράστιες, θα πρέπει να μειωθεί να μειωθούν. Επομένως η συνεργασία έχει σαν στόχο να καταλήξει σε μία μείωση κατά 70% της νησιμότητας ε, της ασθένειας αυτής με το 2020. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Τώρα, η προτεραιότητα για τις έρευνες για τον καρκίνο. Χρειάζεται μια, ένας καλύτερος συντονισμός και θα πρέπει να συγκρίνουμε τις επιδόσεις. Δηλαδή και τις, την ενημέρωση και τα στοιχεία που αφορούν την υγεία. Θα πρέπει να συλλέγουμε τα στοιχεία αυτά, να τα αναλύουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε καλύτερα στην καταπολέμηση τη ασθένεια. Μέχρι το 2003 πρέπει να έχουμε πλήρη στοιχεία που θα αφορούν όλα τα κράτη-μέλη και τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα για πρώτη φορά πλέον. Ε, θα προσπαθώ να είμαι γρήγορη, να είμαι σύντομη. Τώρα οι προτάσει ποιε είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και ε, πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω για να καταπολεμήσει τον καρκίνο. Πρέπει να χρησιμοποιούμε καλύτερα του πόρου που επί του παρόντο είναι πολύ περιορισμένοι και δεν διατίθενται ευρύτερα. Θα πρέπει να προλάβουμε τι επικαλύψει και θα πρέπει να ε, περιορίσουμε τη γραφειοκρατία. Υπενθυμίζω ότι παρά τι σημαντικέ προσπάθειε που έχουν καταβληθεί ο αριθμό των εξετάσεων για, την, για τον εντοπισμό, για την ανείχνευση δεν, έχει, δεν φτάνει μέχρι στιγμή ε, τον ε, ελάχιστο αριθμό που απαιτούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ο αριθμός ε, γίνει, ο αριθμός φτάνει στις ε, στην πρόταση που γίνεται στην ανακοίνωση, τα πράγματα θα βελτιωθούν. Θα πρέπει όμως οι εξετάσει αυτές να αφορούν το 100% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στα πλαίσια αυτη τη συνεργασια μια συγκεκριμένη δομή. Αυτή η δομή θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι υπάρχει μια, μια πρόταση για να δημιουργηθεί ένα φόρουμ, μια ομάδα ε, κατευθυντική με διάφορες ομάδες εργασίας. Ε, θα πρέπει να ε, απλουστεύσουμε τα πράγματα. Θα πρέπει η Κομισιό να μας απαντήσει στο θέμα αυτό. Μετά η Ευρώπη έχει μια χρηματοδότηση για την καταπολέμηση του καρκίνου. Μέσα στα πλαίσια του έκτου πλαισίου, προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και μέσα στα πλαίσια των δύο προκηρύξεων διαγωνισμού στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο υπάρχουν 750.000 ευρώ τα οποία δίδονται για την καταπολέμηση. Εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια ευρώ, συγγνώμη, τα 750 αυτά είναι λίγα, ε, δεν ξέρω. Το πρόβλημα είναι τα χρησιμοποιούμε όμως καλά. Αυτά δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι ερωτήσεις ε, που θέτουμε κύριε Πρόεδρε. Προσπαθώ να ήμουν σύντομη και ελπίζω να ήμουν και αρκετά σαφής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκροστέτ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είχαν αρκετή πειθαρχία οι συνάδελφοι στα πρώτα σημεία της μέσης διάταξης και αυτοί οι οποίοι μένουν πληρώνουν το τίμημα αυτής της έλλειψης πειθαρχίας. Ίσως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί για την τήρηση των κανόνων. Τρεις ομιλητές και πάλι σας παρακαλώ να βοηθήσετε για να μπορούμε να τελειώσουμε πιο γρήγορα. Ο κύριος Χατζημαρκάκης πρώτος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και από τη δική μας ομάδα να χαιρετήσω αυτή την πρωτοβουλία. Θέλω να ευχαριστήσω την συγγέντρια για αυτά που είπε. Οι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήδη είναι ενεργοί εδώ και πολύ καιρό για τον, στον αγώνα κατά του καρκίνου. Υπήρξαν διάφορε διαπαραταξιακέ ομάδε. Υπάρχει ομάδα Ευρωβουλευτέ εναντίον του καρκίνου και υπάρχουν επίση πρωτοβουλίε έρευνα που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και οι οποίε είναι καλόδεκτε. Στι 12 Νοεμβρίου Συζητήσαμε ήδη για μια άλλη ασθένεια με αντίστοιχο αντίκτυπο για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, Αλσχάιμερ και δεν θυμάμαι ποια άλλη αρρώστια. Και ξέρουμε περισσότερα για το Αλσχάιμερ από ότι για τον καρκίνο. Ξέρουμε ότι μια υγιής, ένα, υγιής, ένα υγιές σχήμα ζωής βοηθάει να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση και το ίδιο ισχύει και τον καρκίνο. Χρειάζεται μια ένα υγιή τρόπο ζωή. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε τι πληροφοριακέ εκστρατείε προ του πολίτε. Και επίση, και όπω και στην περίπτωση του Αλτσχάιμερ, προσκρούμε στην ε, στον τομέα της έρευνας σε πολλή γραφειοκρατία και πολλή επικάλυψη προσπαθειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτή τη γραφειοκρατία και να αποφύγουμε τις επικαλύψεις στον τομέα της έρευνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα αποτελέσματα των ερευνών να γίνονται προσβάσιμα σε, όλους, σε όλη την κοινή γνώμη. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παίρνουν κονδύλια θα έχουν την υποχρέωση να δημοσιεύουν και τα πορίσματά τους. Και στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να αναφερθεί και ο τομέας των ευρωπαϊκών τεχνιών. Δεν πρόκειται να συζητήσω αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, αλλά κρατάει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία με τις τεχνίε, Το γνωρίζει και ο πρόεδρος μας, γιατί έχουμε την πρόθεση να κάνουμε και μία ακρόαση. Παραμένει ακόμα σημαντικότερο το θέμα της πρόβλεψης. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε η περιοχή με την καλύτερη πρόληψη στον τομέα του καρκίνου και δεν χρειάζεται να περιμένουμε, όπως λέει η κυρία Γκροστέτ, μέχρι το 2013. Μπορούμε ήδη να ζητήσουμε από το νέο επίτροπο που προέρχεται από τη Μάλτα να προχωρήσει σε σχέση με αυτές τις δράσεις πρόληψης. Ο κύριος Κορέα Δικάμπους. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή είναι χρήσιμη, αλλά είναι ελλειπής και ανεπαρκής. Γιατί, σας το λέω αυτό, είναι χρήσιμη γιατί συλλέγει και ενσωματώνει σε ένα έγγραφο όλες τις πολύ λογικές συστάσεις και τις πολύ ρεαλιστικές συστάσεις σε ό,τι αφορά τον αγώνα κατά του καρκίνου, συγκεκριμένα μια σειρά στόχων κτλ. Αντίθετα με ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν, τώρα έχουμε σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους. Όλοι συμφωνούμε λοιπόν με αυτήν την ε, αντιμετώπιση και την πρόωρη ανείχνευση του καρκίνου του παχαίου σεντέρου, της, του τραχύλου της μήτρας και του στήθους σε ό,τι αφορά τις, ε, τους πρακτικούς κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούνται, αγώνες κατά των διακρίσεων, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα πλαίσιο υπαριθμών 7 για να υπάρξει μεγαλύτερη έρευνα στον τομέα αυτό και να κατευθύνουμε καλύτερα τις ε, έρευνες στον τομέα αυτό και ιδίως τα μητρώα πληροφόρησης, αυτά είναι εκεί που μπορεί να προκύψει η μεγαλύτερη προσθέμενη αξία σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του καρκίνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι πληροφορίες που βρίσκονται στα εθνικά και περιφερειακά μητρώα. Η πρόταση όμως είναι ιδιαίτερα εύθραυστη. Προτείνεται μια εταιρική σχέση με στόχους οι οποίοι είναι ασαφείς, χωρίς να έχει μια οργανική σύνδεση το σύνολο των μέτρων και χωρίς καμία χρηματοδότηση πέραν αυτής της χρηματοδότησης που υπάρχει ήδη. Δεν προβλέπει καμία νέα οργανωμένη δράση αυτή η πρόταση λοιπόν και έχουμε να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη πόρων. Προφανώς οργανώνει καλύτερα τις ε, δυνατότητες που υπάρχουν τώρα, αλλά είναι <clears throat> πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από μια νέα πρόταση. Εγώ δεν νομίζω ότι λείπουν δυνατότητε να έχουμε εναλλακτικέ λύσει. Η Κομισιόν μπορεί να χρησιμοποιήσει το κέντρο για τον έλεγχο των ασθενειών για να περιλάβει και ασθένειε, οι οποίε δεν είναι μεταδοτικέ για να αντιμετωπίσει τη δυνατότητα να οργανώσει τη συλλογή πληροφοριών για ασθένειε, οι οποίε δεν είναι ε, μεταδοτικές μεταξύ των οποίων και ο καρκίνο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταχύτατη απάντηση από την Κομισιόν, κύριε Μπότακ. Μπότακ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συζητεί την ανακοίνωση αυτή και στις 29 Σεπτεμβρίου ήταν παρόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ημέρα που έγινε η ανακοίνωση αυτή και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Ε, τέθησαν ορισμένα ερωτήματα που θα ήθελα να προσπαθήσω να απαντήσω. Πρώτο ερώτημα σχετικά με τη δομή. Η πρότασή μας είναι να δημιουργήσουμε μια εταιρική σχέση η οποία θα εντάσσεται σε στο πλαίσιο κοινών δράσεων από του χρόνου και μετά μέχρι το 2013 ζητήσαμε να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος ή ενδιαφερόμενοι αυτό έγινε και θα γίνει την επόμενη εβδομάδα η πρώτη συνάντηση για τη δημιουργία αυτής της εταιρικής σχέσης την επόμενη τρίτη και η συμφωνία για τη δομή αυτής της εταιρική σχέσης θα λάβει χώρα σε αυτή τη συνεδρία. Οι ίδιοι συμμετέχοντες θα αποφασίσουν για τη δομή. Επίσης προσπαθήσαμε να εντάξουμε και άλλα ε, στοιχεία, παραδείγματος χάρη εικονική συμμετοχή ε, μέσα στο πρόγραμμά μας δηλαδή αυτοί που θέλουν να συμμετάσχουν αλλά δεν μπορούν να μπορούν να λάβουν μέρος και να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και ε, ε, επίσης ε, θα προσπαθήσουμε ενέργειες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να τις επαναφέρουμε στο τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και τα περισσότερα κράτη-μέλη μπορώ να σας πω ήδη από τώρα ότι αντέδρασαν θετικά και τους περιμένουν, τα περιμένουμε να έρθουν και στη συνεδρία στην επόμενη εβδομάδα τώρα για την πρόληψη Συμφωνώ ότι η πρόληψη και η γύρινη ζωή είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία και βοηθούν. Ήταν ψηλή, ε, τα πρώτη προτεραιότητα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πρόληψη ε, για το αλκοόλ, για την ε, άσκηση για την απαγόρευση του καπνίσματος ήταν πρωτοπόρος η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά τα και παρόλο που οι στόχοι είναι μετριοπαθείς ελπίζουμε η δουλειά που κάνουμε τώρα και που θα οργανώσουμε την επόμενη εβδομάδα και για τα επόμενα τρία χρόνια να αποδώσει περισσότερους καρπούς Σίγουρα εάν λείπει κάτι από την πρότασή μας θα μας ε, το υπενθυμίσουν οι ενδιαφερόμενοι. Ε, ο συνάδελφός από την έρευνα μπορεί να πάρει το λόγο λέει ο πρόεδρος αλλά πολύ σύντομα ναι ευχαριστώ πρόεδρε να συμπληρώσω για το τομέα της έρευνας σίγουρα χρειάζεται καλύτερο συντονισμός ερευνητικών προσπαθειών και ο στόχος του να, να υπάρξει συντονισμός για όλη την έρευνα που γίνεται μέχρι το 2013 είναι πολύ φιλόδοξος η, σίγουρα στην ε, έγινε πρόσβατα η μεγαλύτερη δυνατή διαβούλευση που έχει γίνει ποτέ για θέματα καρκίνου και όπου έγινε η διαβούλευση για την έρευνα και θα αποφασίστηκε να χρηματοδοτηθεί ένα δίκτυο ε, συντονισμού της έρευνας για το καρκίνο στην Ευρώπη ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι τι άλλο στο οποίο θα διαθέσουμε 12 εκατομμύρια ευρώ είναι τα κέντρα αριστείας για το θέμα του καρκίνου και κάποια άλλα κέντρα γενικότερα για τον καρκίνο. Θα χρηματοδοτήσουμε λοιπόν και τα, όλα τα κέντρα αυτά ελπίζουμε και επίσης θα επικεντρωθούμε με άλλα 12 δις ε, ευρώ για τον παιδικό καρκίνο παιδιατρικό καρκίνο. Ευχαριστώ η συγγετρία κυρία Γκροστέτ. Θέλει να ξαναπάρει το λόγο ή όχι. 30 ε, δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε. Σα διαβεβαιώνω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου που πήραν το λόγο. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα ύψη τη σημασία μείζον θέμα. Θα πρέπει τελικά να καταλήξουμε σε μια κατάσταση ε, και αυτό είναι ο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου τα κράτη-μέλη θα δεσμευθούν. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει κάποια χρήματα, τα οποία όμως να μην χρηματοδοτήσουν κάποιες συναντήσεις και συνεδριάσεις. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί στο συντονισμό που θα κάνουμε πάνω χάρη για την έρευνα. Ε, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους συναδέλφους και αν έχουν καλές προτάσεις ε, εδώ ε, να κάνουν, ε, είμαι στη διάθεσή τους. Ευχαριστώ πολύ. 28 Ιανουαρίου, 2 Φεβρουαρίου θα είναι η προθεσμία της τροπολογίας. Μπορούν να μας δώσουν 5-10 λεπτά ακόμα οι διερμηνείς. Μπορούμε τότε να αντιμετωπίσουμε το θέμα του κ. Μπίτικοφερ. Γίνεται. Κύριε Μπίτικοφερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή η Οικονομική είναι η επί της ουσίας αρμόδια Επιτροπή για την ε, πολιτική ανταγωνισμού και εμείς δίνουμε απλώς μια γρομοδότηση. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω τρία βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να ενδιαφέρουν τη δική μας Επιτροπή. Καταρχήν το θέμα πώς την τωρινή χρηματοοικονομική και οικονομική κρίση μπορούν οι εθνικές ενισχύσεις να επηρεάσουν το τομέα του ανταγωνισμού. Δεύτερον, πώς αυτή η οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τρίτον, τι θα πρέπει να κάνει η ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού για να τονώσει την καινοτομία στην ευρωπαϊκή, στον ευρωπαϊκό τομέα. Συνθηματολογικά και μονάχα θα σας αναφέρω τα σημεία τα οποία κατά τη δική μου άποψη θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην γνωμοδότηση της Επιτροπής μας. Η Κομισιόν έχει, και χαίρομαι γι' αυτό, στην έκθεσή της για τον ανταγωνισμό, περιλάβει ένα κεφάλαιο για τα καρτέλ και τους καταναλωτές. Εγώ νομίζω ότι είναι απαραίτητο μέσα σε μια έκθεση για ανταγωνισμό να έχουμε και ένα κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιπλέον. Δεύτερον, πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και όχι μονάχα στους original equipment manufacturers αλλά και στη σχέση μεταξύ εταιριών και ε, υπεργολάβων και τροφοδότων. Τρίτον, θέλουμε να εξασφαλίσουμε τον τομέα της ε, πληροφορίας όπου υπάρχει όλο και μεγαλύτερη, μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Τέταρτον, η Κομισιόν έχει κάνει πολλά με, και θα έκανε ίσως και περισσότερα με την υποστήριξη των 100 μελών για τον ανταγωνισμό στον τομέα των δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού μάλλον, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη και τις συνέπειες που προέρχονται από τον ανταγωνισμό στην, μετά από τα συμπεράσματα της διάσκεψης της Κοπενχάγης για την κλιματική αλλαγή. Τέλος, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών τίθεται το θέμα του πώς οι Ευρωπαίοι ρυθμιστές οι ρυθμιστικές αρχές λοιπόν στον τομέα των τηλεπικοινωνιών μπορούν να αποτελέσουν ένα φορέα ο οποίο θα εξασφαλίσει ανεξάρτητα τον ανταγωνισμό στον τομέα αυτό. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν επομένως να μπορέσουμε εμείς να συμβάλλουμε στο θέμα αυτό στην έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών για το ποιες θα ήταν οι πιο πρόσφερες στρατηγικές οι οποίες θα επιτρέψουν και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παίξουν κάποιο ρόλο. Αυτά τα σημεία τα οποία έχω καταγράψει ω ενδιαφέροντα για την Επιτροπή μας θα ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων αν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προβληματική. Έχουμε το πρόβλημα βέβαια ότι θα είμαστε σε πίεση χρόνου λόγω των ακροάσεων των Επιτρόπων. Παρακαλώ τον κύριο Μπιτικόφερ και τους σκιώδεις εισηγητές να βρουν κάποιο τρόπο ώστε εν συντομία, εν ταχυτή